Uh, Συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, έχω την χαρά σήμερα να προεδρεύω αυτή της ακρόασης για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Σας καλωσορίζω θερμά όλους και ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους μας. Ξέρετε ότι τον Απρίλιο του 2018 η Κομισιόν υπέβαλε το λεγόμενο πακέτο για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, που αποτελείται από έναν κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολής Στοιχείων και Διατήρηση Στοιχείων. Μια οδηγία για, το, για τη θέσπιση εναρμοσμένων κανόνων για τον διορισμό των νόμιμων εκπροσώπων για το σκοπό της συλλογή υποδεικτικών στοιχείων σε ποινικέ υποθέσεις. Ο κανονισμός που και όχι η οδηγία που σημαίνει ότι ισχύει άμεσα χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί ε, στο εθνικό δίκαιο δημιουργεί μια ευρωπαϊκή εντολή υποβολή στοιχείων που επιτρέπει σε δικαστική αρχή σε ένα κράτος μέλος να λαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία όπω email, μηνύματα κειμένου σε εφαρμογές και άλλε πληροφορίε για να προσδιορίζει την ταυτότητα ενό δράστη ω πρώτο βήμα άμεσα από τον πάροχο υπηρεσιών ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε άλλο κράτο μέλο, χωρίς το άλλο κράτος μέλος να ενημερώνεται ή να συμμετέχει στη διαδικασία ο οποίος με τη σειρά του θα υποχρεούται να απαντά εντός 10 ημερών και εντός 6 ώρων σε περίπτωση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δημιουργεί επίσης μια ευρωπαϊκή εντολή ε, διατήρηση στοιχείων που επιτρέπει σε δικαστική αρχή ενός κράτους μέλους να ζητά από πάροχο υπηρεσιών ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε άλλο κράτος μέλων να διατηρεί συγκεκριμένα δεδομένα χωρίς το άλλο κράτος μέλος να ενημερώνεται ή να συμμετέχει προκειμένου να μπορούν αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω της ε, δικαστικής, αμοιβές δικαστικής συνδρομής μέσω ευρωπαϊκής έλλειψης διερεύνησης ή ε, εντολής σε υποβολή στοιχείων. Η οδηγία αυτή συμπληρώνει το πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός καθώς εισάγει την απέτηση να ορίζεται εκπρόσωπος για τους παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Περισσότερες από τις συζητήσεις αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στον κανονισμό και η Αυστρική Προεδρία ε, στοχεύει στο να καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση. Στο Κοινοβούλιο έχουν γίνει διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις λόγω της περιπλοκότητας του ζητήματος και εδώ στο, στην Επιτροπή μας έχουμε παρακολουθήσει το ζήτημα από κοντά. Η Κομισιόν έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το νέο σύστημα θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε οι αρχές επιβουλής του νόμου και οι δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για τις έρευνές τους, για τη δίωξη και την καταδίκη εγκληματιών και τρομοκρατών. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες ε, ε, και άλλοι ειδικοί ε, καθώς και εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ε, θέσει και εκφράσει μια σειρά από ανησυχίες που έχουν όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που προσφέρει, προσφέρει αυτός ο μηχανισμός, ε, την διαλειτουργικότητα και τις επιπτώσεις σε άλλα συστήματα, την αναλογικότητα, την έλλειψη εναρμόνισης των εθνικών συνταγματικών προδιαγραφών, μεταξύ πολλών άλλων. Λόγω λοιπόν της σημασίας του ισχύοντος συστήματος και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει το νέο προτινόμενο σύστημα είναι πολύ σημαντικό να διοργανώσουμε σήμερα μια δημόσια ακρόαση όπου θα συμμετέχουν διάφοροι επαγγελματίες, πάροχοι, εμπειρογνώμονες στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων για να σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα. Στην εποχή λοιπόν της σύγχρονης τεχνολογίας ε, αναδύονται νέα ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και τους περιορισμούς της τεχνολογίας. Γνωρίζουμε ότι το θέμα των ηλεκτρονικών στοιχείων ε, τέμνει μια σειρά από ζητήματα όπως είναι νέες τεχνολογίες, επιβολή του νόμου και τον κίνδυνο του αποκαλούμενου διαφανούς πολίτη. Θέμα που έχει αναδείξει με αποφάσεις του και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και που έχει συζητηθεί και στο πλαίσιο ε, άλλων θεμάτων όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα πράγματα, δεν θα το κάνω όμως. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, για να τοποθετηθεί, γιατί έχουμε και εξαίρετους προσκεκλημένους σήμερα που θα μπορέσουν να φωτίσουν το θέμα αυτό ε, με έναν εξαιρετικά ολοκληρωμένο τρόπο. Τους ε, καλωσορίζω. Τρία πάνελ θα γίνουν, όπως αναφέρεται και στη μίληση διάταξη. Κάθε πάνελ, θα, κάθε ομιλητής μάλλον, θα έχει το λόγο για 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα γίνονται ερωταπαντήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, που είναι η Birgit Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε έμπειρη συγκήτρια σε αυτό το θέμα που όπως είπαμε είναι πραγματικά μια νέα πρόταση, μια νέα δέσμη προτάσεων αυτή της Κομισιόν Ριξικέλευτη. Μπίργκετ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Κλοντ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μου χαρά και πραγματικά προσβλέπω στις απόψεις και τα στοιχεία που θα ακούσουμε σήμερα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας για αυτήν την δέσμη μέτρων για τα ηλεκτρονικά παιδευτικά στοιχεία. Για τους σκιώδεις συναδέλφους μου, αλλά και για τους άλλους ευρωβουλευτές που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, η ακρόαση αυτή θα μας βοηθήσει ώστε να συλλέξουμε σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο των σημαντικών τοποθετήσεων, προβληματισμών, ανησυχιών που έχουν εκφραστεί γύρω από τις νέες αυτές εντολές υποβολής στοιχείων και διατήρησης στοιχείων. Και χαίρομαι και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις προτάσεις ε, για τους ομιλητές που έλαβα από τους ε, συναδέλφους μου. Δεν είναι η πρώτη ακρόαση που διοργανώνουμε για την πρόταση της Κομισιόν. Αντιθέτως, έχουμε ήδη διεξαγάγει μια σειρά από εσωτερικές συναντήσεις και συνεδριάσεις με ε, την Κομισιόν, με εμπειρογνώμονες στον τομέα της προστασίας των ε, πολιτικών, των προσωπικών ε, δεδομένων και πολλούς άλλους και είμαι βέβαιο ότι όχι μόνο εγώ αλλά και οι άλλοι σκιώδεις έχουν προβεί και σε μια σειρά από άλλους, άλλες διμερείς επαφές με εισαγγελίε, αστυνομικές αρχές κτλ. Η εντολή αποβολή και διατήρηση στοιχείων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της ε, συνεργασίας ε, των δικαστικών και αστυνομικών αρχών και θα ε, βοηθήσει το συνολικό περιβάλλον. Λόγω της, της δικημενόμενης φύσης των ε, ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων ε, είναι λογική η πρόθεση της Κομισιόν να επιταχύνει και να ενισχύσει τη συνεργασία. Όμως η πρόταση αυτή αποτελεί πραγματικά καινοτομία όσον αφορά την ε, διασυνορική συνεργασία στο ποινικό δίκαιο. Και ενώ τα εργαλεία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ε, μέχρι σήμερα είχαν τον ε, χαρακτήρα ε, διμερού, διμερών επαφών, το σχέδιο κανονισμού για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία προτείνει την αναγνώριση, την αυτόματη αναγνώριση εντολών από παρόχους υπηρεσιών, ακόμα και αν αυτές οι εντολές προέρχονται από άλλο κράτος μέλος. Το, οι αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενημερώνονται μόνο αν ο πάροχος ε, υπηρεσιών του κράτους μέλους ε, ε, αυτού δεν απαντά, δεν ανταποκρίνεται στην εντολή. Αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με την ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και λόγω της ευαισθησίας της φύσης της συνεργασίας στον δικαστικό τομέα υπάρχουν ακόμη και ανησυχίες και αμφιβολίες για τη νομική βάση του κανονισμού. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι αρχέ επιβολή των νόμων και την ε, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εμπλεκομένων. Η πρόταση προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των εντολών υποβολής και διατήρησης στοιχείων ε, από παρόχους υπηρεσιών που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και επιδεδομένων περιεχομένου τα metadata. Ακόμα και με τα metadata όμως, με τα μεταδεδομένα, μπορεί κανείς να σχηματίσει μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή κάποιου ανθρώπου, με ποιον συναντιέται, που κινείται, σε ποιους χώρους, τι του αρέσει να διαβάζει, τι ψάχνει στο ίντερνετ και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό η επιτάχυνση της συνεργασίας μέσω τέτοιου είδους ε, σύντομων δρόμων πρέπει να συνοδεύεται από μεγάλη προσοχή, ώστε αυτά τα νέα καθεστώτα να μην αντίκυνται στις βασικές και θεμελιώδεις μας αρχές. Ελπίζω λοιπόν η σημερινή ακρόαση να φωτίσει το θέμα, ιδίως από την άποψη της πρακτικής ανάγκης αυτού του νέου εργαλείου, να φωτίσει το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων εργαλείων και την αναλογικότητα ε, στο βαθμό που αυτό αυτή χαρακτηρίζει τη νέα ε, πρόταση, καθώς και ορισμένα νομικά ζητήματα, ποινικέ διατάξεις των συνθήκων, ε, τους χάρτες ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και προστασίας προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και με την εξεδαφική επιβολή του νόμου, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικονομικές εγγυήσεις, την απουσία ε, κοινών προτύπων, αλλά και πρακτικά θέματα, όπως για παράδειγμα την ικανότητα ενός παρόχου υπηρεσιών να ελέγχουν την γνησιότητα ή και την, ε, τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των εντολών που θα λαμβάνουν. Ελπίζω λοιπόν να συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ενημερωμένη ε, απόφαση να δώσω το λόγο στον καθηγητή Δ. και από το Πανεπιστήμιο της Βόνης ε, για να μας παρουσιάσετε τη μελέτη και μια αξιολόγηση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια, πιστηρία. Από το τμήμα πολιτικής ε, κατόπιν αίτημα της δικής μας Επιτροπής. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα απορίσματα τη έρευνα μα στα 10 λεπτά. Είναι φιλόδοξο ο στόχο, αλλά σα υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι παίρνει το χέρι μου. Η παρουσίασή μου θα είναι σε τρία τμήματα. Ένα τμήμα για την ουσία τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια. Κατά δεύτερον, για την προστιθέμενη αξία και τα μειονεκτήματα τη πρόταση. Και θα κλείσω με κάποια πορίσματα για εναλλακτικέ λύσει και για το μέλλον για το πεδίο εφαρμογή και το περιεχόμενο τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια δωρά. Παρά τον γενικό όρο ηλεκτρονικά τεκμήρια, περιορίζεται η πρόταση σε δεδομένα τα οποία φυλάσσονται από παρόχους. Η πρόταση λοιπόν αντικαθιστά το πρόγραμμα διαστοριακής συνεργασίας ε, μεταξύ των αρχών ε, των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι προτάσεις λοιπόν περιλαμβάνουν δύο νέα εργαλεία συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολή Στοιχείων και διατήρηση στοιχείων. Σύμφωνα με τον ε, νομοθεσία του κράτους που υποβάλλει την, το αίτημα αν ο πάροχος λοιπόν δεν δεν ε, ανταποκριθεί στις υποχρεάσεις τους, υποχρεούται από το κράτος μέλος εκτέλεσης να το πράξει. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Υποβολή Στοιχείων και το νέο καθεστώς υποδεικνύει ότι το δεύτερο κράτος μέλος θα υποχρεούνται μόνο εφόσον αρνηθεί να συνεργαστεί ο πάροχος. Ένα δεύτερο θέμα. Ποια είναι η προσθέμενη αξία του νέου αυτού καθεστώτος σε σύγκριση με το τρέχον πλαίσιο αυξάνει την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ηλεκτρονικά δεδομένα, δημιουργώντας νέους μηχανισμούς άμεσης συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβόλης του νόμου και των παρόχων και έτσι θα μας γλιτώσει σε βάθος χρόνου και πόρους και χρόνο η νέα πρόταση. Το νέο πλαίσιο, ωστόσο, δεν θα ξεπεράσει τον καταγερματισμό και την ε, διαφορετικότητα που υπάρχει στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την, ε, τον τρόπο τήρησης και παραγωγής τέτοιων δεδομένων. Καταρχάς, η διατήρηση τέτοιων δεδομένων θα παραμείνει στα χέρια των εθνικών κρατών μελών. Δεν θα αλλάξει τίποτα εδώ. Κατά δεύτερον, το προτινόμενο καθεστώ διασυνοριακή συνεργασία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην νομοθεσία του κράτου μέλου που υποβάλλει την εντολή. Και σε κάποιο βαθμό, όπω ε, σε ό,τι αφορά την ασυλία και τα προνόμια, στο καθεστώ, στο νομοθετικό καθεστώ, του κράτου μέλου που δέχεται την εντολή. Άρα δεν υπάρχει ένα αρμονισμένο πλαίσιο για το πώ χορηγούνται τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι τώρα τα μειονεκτήματα. Θα ήθελα να τονίσω δύο βασικέ ανησυχίε μα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση και την δικαιοδοσία και το δεύτερο στοιχείο σε ό,τι αφορά την προστασία των, των θεμελιδών δικαιωμάτων και την ε, διάμεση αναθεώρηση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επεκτείνει το παιδί εφαρμογή και σε παρόχους που έχουν έντρα και φυλάσσουν τα τεκμήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν έχει επιπτώσεις και στο διεθνέ επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών. Ε, κοιτάζοντας λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι προτάσεις αυτές ε, θα είναι σε συνάρτηση με το διεθνέ δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το πλαίσιο τη διεθνού συνεργασία με τρίτα κράτη και να προκαλέσει και ζητήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της δικαιοδοσίας. Επίσης, οι αντικρουόμενες υποχρεώσεις για τους παρόχους για να παρέχουν ή να μην παρέχουν, να υποβάλλουν ή να μην υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά, ενδεχομένως να προκαλέσουν αβεβαιότητα και στους παρόχους και στους χρήστες. Εντός της Ένωσης τώρα η άμεση συνεργασία θα επηρεάσει την περιφερειακή κυριαρχία των ε, κρατών στο οποίο βρίσκεται ο πάροχος των υπηρεσιών. Το νέο καθεστώς αγνοεί λοιπόν την ευθύνη του κράτους μέλους εφαρμογής σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της επικρατείας τους. Κοιτώντας το θέμα λοιπόν της περιφερειακής επικυριαρχίας, η νέα πρόταση πάει πολύ παραπέρα σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση και υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά το άρθρο 82 παράγραφος 1 και κατά πόσον αποτελεί μια ικανοποιητική νομική βάση για την διάταξη αυτή. Δεύτερο σημείο σε ό,τι αφορά την τα θεμελιώδη δικαιώματα και την δικαστική αναθεώρηση. Δεν προβλέπεται επαρκείς ε, δικλείτες ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αποστρεί από το άτομο προσφυγή σε δικαστικές αρχές ε, και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρελευάσει περιλάμβει και κάποιες διτάξει για την προστασία της ασφάλεια και η πρόταση δημιουργεί υποχρέωση τα δεδομένα περιεχομένου και συναλλαγών να χορηγούνται ακόμα και αν δεν πληρούνται οι όροι του κράτους μέλους εφαρμογής και έτσι το νέο καθεστώς ουσιαστικά ε, υπονομεύει ένα καθεστώς προστασίας σε ό,τι αφορά τη χώρα όπου εκτελείται η εντολή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο βαθμό που καλύπτονται αυτά από την πρόταση, η προστατευτική αυτή λειτουργία δεν ασκείται από τα κράτη-μέλη στην ε, επικράτη της οποίας εκτελείται η εντολή, αλλά από τον πάροχο ή από την χώρα που εκδίδει το ένταλμα. Κανένα από του δύο όμω δεν είναι αρμόδιο για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην επικράτεια του κράτου μέλου υποδοχή. Υπάρχει λοιπόν μια μετατόπιση των ε, αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων σε ό,τι αφορά την ευθύνη αυτή από το κράτος μέλος ε, υποβολής στο κράτο μέλο υποδοχή του, της Η πρόταση δεν προβλέπει το δικαίωμα α, ε, καταγγελίας του αιτήματο σε δικαστήριο της χώρας. Δεν μπορούμε λοιπόν να γίνεται για διαδικασία στο ίδιο το κράτος υποδοχής του αιτήματο. Οι πάροχοι τώρα έχουν νομικά μέσα στη διάθεσή τους, ανώμα μέσα στη διάθεσή τους, στη χώρα Υποδοχή του αιτήματο, αλλά ενδεχομένω το, το μάλλον ο πάροχο δεν μπορεί να υποβάλει τέτοια αγωγή στο κράτος μέλος υποβολή του αιτήματο, παρά το γεγονό ότι δικοί του κανόνες εφαρμόζονται. Τελευταίο σημείο τώρα για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα μειονεκτήματα που περιλαμβάνει η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου σε τι βαθμό θα μπορούσε να παρατελέσει εναλλακτική λύση μια αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εντολής Ερευνών. Η πρόσβαση σε γρήγορα στοιχεία βασικά βασίζεται στην ε, κατάργηση εμποδίων και στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό ήταν υπερβολικό διακύβευμα για την συνεργασία. Ύστερα, θα πρέπει να υπάρχει και διμερείς συμφωνίες σε ό,τι αφορά την πραγματεύσεις για τα ε, ενδιάμεσα πρωτόκολλα ή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ετρεσε των ε, παροχών ή μονομερείς εφαρμογές ε, δικαιοδησίας. θα πρέπει να είναι αυστηρός περιορισμένες για να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των χωρών και μεταξύ των παρόχων στο βαθμό του δυνατού. Τρίτον, τα κράτος μέλος εφαρμογής θα πρέπει να συμμετέχει και στην έκδοση της ε, εντολής. Για παράδειγμα, στα, σε άλλα συστήματα υπάρχει ένα σύστημα κοινοποίηση τη εντολή προκειμένου να αναλάβει την έκδοση του αιτήματο στην επικρατεία του κράτου υποδοχή. Τέταρτον, τα υψηλά πρότυπα προστασία που καθορίστηκαν στο χώρο δικαιοσύνη και συνεργασία εφαρμόζονται από το κράτο μέλο σε υποδοχή τη εφαρμογή. Και ιδιαίτερα στα δεδομένα αυτά, τα τεκμήρια αυτά θα πρέπει να διατηρούνται. τέλο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται αποτελεσματική δικαστική αναθεώρηση και στα δύο κρατημέλη και σε αυτό τη έκδοση τη εντολή και σε αυτό τη υποδοχή τη εντολή. Και επίση θα πρέπει να υπάρχουν έντομα μέσα για να καταγγελθεί η νομιμότητα τη εντολή στο κράτο μέλο υποβολή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Και τώρα να περάσουμε στην πρώτη, στο πρώτο γύρο. Θα ακούσουμε τις εμπειρίες των εμπλεκομένων φορέων. Ο καθηγητής Δ. θα πρέπει να φύγει σύντομα. Αν έχετε λοιπόν ερωτήσεις για την ε, έρευνα, η Σοφή και μετά η Μπρικίτ, η εισηγητρία, η να ακούσουν πρώτα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση της μελέτης. φοβούμαι ότι δεν είμαστε και τόσο καθυσυχασμένοι ότι όλα πάνε καλά με αυτή την πρόταση. Κάναμε διάφορες, είχαμε διάφορε ανησυχίε και εσεί στην ουσία τι επιβεβαιώσατε. Ερώτησή μου είναι γιατί εγώ δεν είμαι κατηγορηματικά αντίθετη στην ιδέα. Αν πραγματικά μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά οι προστασίε θα πρέπει επίση να είναι εξασφαλισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για την ώρα, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, που δεν είναι η μόνη νομική προστασία που χρειάζεται, σε πολλά κράτη-μέλη καλύπτεται ακόμα από την απόφαση του Συμβουλίου του 2008. Γιατί η αποκαλούμενη οδηγία της αστυνομίας δεν έχει εφαρμοστεί. Οπότε, ακόμα και αν εφαρμοστεί πλήρω η οδηγία της αστυνομία σε όλα τα κατημέλη, είναι αρκετή ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε η Κομισιόν να έχει συνοδέψει αυτή την πρόταση με μια πρόταση για κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Τρίτη ερώτηση. Τι άλλα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις και οι ανησυχίες που τονίσατε εσείς. Και τελική μου ερώτηση είναι δεν πρόκειται μόνο για ηλεκτρονικές αποδείξεις εντός της Ένωσης, πρόκειται και για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, που κατά μένα είναι απαράδεκτο να δώσουμε σε μια τρίτη χώρα άμεση πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούσαμε και να σχίσουμε και το GDPR, άμα είναι έτσι. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας φωτίσετε και γι' αυτό. Είναι μια ερώτηση η οποία προέκυψε και στις συζητήσεις με τους ε, ε, πρέσβεις των ΗΠΑ. Ακούσουμε ακόμα δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ σύντομα. Η ε, Μπίργκιτ. Ευχαριστώ. και εγώ Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη μετά την παρέμβαση της συναδέλφου της κυρίας Σοφίντφελντ αναφέρατε ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κατά πόσον το ευρωπαϊκό ένταλμα ερευνών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον ελεκτικό μοντέλο. Μου είχε προκαλέσει έκπληξη γιατί τα χρονικά περιθώρια τα οποία δίνουμε σε μία αρχή για να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα είναι τώρα πιο μεγάλα, ενώ οι πάροχοι τώρα καλύτερα να απαντήσουν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό δεν ξέρω αν είσαστε σωστό άνθρωπο να το ρωτήσω αυτό, αλλά θα μας, μπορούσατε να μα πείτε κατά πόσον θα μπορούσατε να φανταστείτε και τα χρονικά περιθώρια στην ε, εντολή έρευνας να γίνουν πιο σύντομα σημαντικά, πιο σύντομα. Ευχαριστούμε η κυρία Κινίτσι. Σα ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Μπόση για την ανάλυση του που πρέπει να πω σε μεγάλο μέρος με βρίσκει σύμφωνη γιατί τόνισε ε, κάποιους και από τους δικούς μας προβληματισμούς. Αν και εγώ πιστεύω πως ε, η ιδέα της ηλεκτρονικής απόδειξης είναι σίγουρα μια ιδέα επί της θα πρέπει να δουλέψουμε με βάση τις απαιτήσει που ε, προκύπτουν στις έρευνες διασυνοριακής φύσης. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στο τελευταίο σημείο που θίξατε και που αφορά τη διαδικασία επανεξέτασης που ορίζεται από το άρθρο 15 του κανονισμού για την ε, υποχρέωση υποβολής και προβλέπει έλεγχο από το κράτος εκτέλεσης τη στιγμή που Ε, υπάρχουν ε, αντιθέσεις ε, με το εφαρμοστέο δίκαιο σε κάποια χώρα ανάλογα με την υπόθεση. Πρόκειται για μια αξιολόγηση που καταρχάς νομίζω μπορούμε να συμμεριστούμε. Όμως μπορεί να είναι δύσκολη στην εφαρμογή της από πλευράς μιας δικαστικής αρχής γιατί δεν υπάρχουν απαιτήσει διοικητικού τύπου. Θεωρείτε λοιπόν πως μια τέτοια αξιολόγηση είναι σύμφωνη με την, ε, το σεβασμό της αρχής της διεθνούς ε, εντολής. Ευχαριστώ. Καθηγητά Μπόσε. Θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Ανέφερα νομικές ε, καλύψεις για τον πάροχο υπηρεσιών. Και εσείς αναφέρετε ε, μία περίσταση όπου η νομική κάλυψη ε, για τον πάροχο της υπηρεσίας χορηγείται από το κράτος έκδοσης. Δεν υπάρχει κάποια γενική νομική κάλυψη για τον πάροχο της υπηρεσίας. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις, οι διατάξεις είναι αρκετά λεπτομερείς. και για να το πω πολύ σύντομα, δεν νομίζω πως εδώ μπορούμε να επικρίνουμε πολλά. Η Κομισιόν προσπάθησε να ε, συντάξει μια ισορροπημένη διατύπωση, λαμβάνοντας υπόψη το, ε, την ε, επιβολή του νόμου και το συμφέρον του παρόχου, από την άλλη. Δηλαδή, σε αυτό δεν θα, δεν θα επέμενα ιδιαίτερα στις επικρίσεις μου. Οι επικρίσεις μου αφορούν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μόνο στοιχείο, ένα σημείο χώρο που προβλέπονται καλύψεις για το κράτος ε, έκδοσης. Χρονικοί περιορισμοί. Για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει κανείς να κατανοήσει ότι σε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Ερεύνης σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι μόνο θέμα της εκτελεστικής αρχής να διαβιβάσει απλά τις πληροφορίες, πρέπει και να τις συλλέξει προηγουμένως. Οπότε έχουμε πάνω κάτω δύο φάσεις και αυτό μπορεί να είναι λόγος για την πρόβλεψη ενός μακρύτερου χρονικού διαστήματος από ότι για έναν ιδιώτη που έχει στην κατοχή του ήδη τις πληροφορίες. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Νομίζω πως ε, στα επόμενα πάνελ υπάρχουν ε, πιο περισσότεροι άνθρωποι της δουλειάς, ας πούμε, της πρακτικής που θα σας απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις σας. Τώρα, η απόφαση του 2008 είναι οδηγία. Το πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό, αλλά εάν μιλάμε για πρόσβαση τα δεδομένα συναλλαγής και ε, περιεχομένου, πιστεύω πως αυτές οι προδιαγραφές δεν είναι ε, αρκετές. Τουλάχιστον από όσα γνωρίζω, ακόμα και η νέα οδηγία δεν περιλαμβάνει καμία διευκρίνηση όσον αφορά ανώτατα εκατότατα τα κατόφλια για τα ερευνητικά μέτρα που στόχο έχουν να συλλέξουν ε, στοιχεία περιεχομένου ή στοιχεία για τις συναλλαγές. Εάν θέλουμε λοιπόν να θεσπίσουμε ομοιόμορφα ευρωπαϊκά στάνταρ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να υιοθετήσουμε μια οδηγία για την εναρμόνιση του νόμου για τις ποινικέ διαδικασίες υπό το άρθρο 82.2 και όχι κανονισμό, μόνο οδηγία. Και υπάρχουν και κάποια άλλα βήματα και προποθέσει που θα πρέπει να τηρηθούν για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μέτρο, αλλά νομίζω αυτό θα ήταν ο μόνο τρόπο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πάντοτε μια μίξη εθνικών κατοφλίων ανάμεσα στο κράτο έκδοση και το κράτο εκτέλεση. Δηλαδή τελικά θα έχουμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ομοιόμορφη προδιαγραφή, τότε αυτό η διπλή θα είναι το μίνιμουμ. Τουλάχιστον εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν θυμάμαι τώρα τη δεύτερη ερώτηση. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Ναι, ήταν τρι, τριπλή η ερώτηση μου και αφορούσε την ολοκλήρωση της προστασίας των δεδομένων και το σχετικό επίπεδο που εν μέρη ήδη απαντήσατε και δεύτερον τι άλλο θα έπρεπε να γίνει για να καλυφθούν ε, οι ελλείψεις και τρίτον η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τι άλλο μπορεί να γίνει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να λάβει απόφαση είτε είναι ναι είτε είναι όχι για τη μεταφορά αυτών των δεδομένων. Αυτή ήταν ε, και η παρατήρησή μου σε σχέση με τις διατάξεις για τη σύμβαση, την εφαρμοστική της συμφωνίας του Σέγγεν για τη διασυνοριακή εποπτεία και την ε, δίωξη. Θα δείτε πολύ λεπτομερείς κανόνες που αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα, την εδαφική ε, κυριαρχία του κράτους όπου αλλοδαπές αρχές εκτελούν μέτρα ερεύνης ή μια σύλληψη ή και προσωρινή σύλληψη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρθρο 89 της Συνθήκης ακολουθεί τελείως διαφορετική νομοθετική διαδικασία από το 82. Οπότε, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Ανέφερα την ε, δικαστική εξέταση. Αυτό ακολουθεί κάπως την διάκριση των ε, καθηκόντων και των εξουσιών ανάμεσα στη, στα κράτη-μέλη. Και νομίζω αυτά είναι τα κυρία ζητήματα. Και βεβαίως, το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλοι παίκτες είναι κατεστημένοι στη ΣΥΠΑ. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ γιατί αλλιώ θα ε, αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν έχω λύση. Υπάρχουν ε, μέτρα Υπάρχουν μέσα. Συγγνώμη. Το MLAD είπε η συνάδελφος, ε, αλλά ας μην γίνει καλύτερα ε, διάλογος. Ναι, λέει ο αλλά ομολογώ ότι δεν έχω λύση από αυτού. Η μελέτη μας επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο ε, στο καθεστώς που ισχύει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και υπάρχουν και αυτές οι πτυχές του θέματος, αλλά δεν τις φωτίσαμε στην ε, μελέτη μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέζε. Και θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και την ε, μελέτη σας. Μπορούμε να πάμε τώρα στην πρώτη μας, ε, στον πρώτο γύρο συζήτησης, εμπειρίες από επαγγελματίες του χώρου με τα υπάρχοντα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλώ τους προσκεκλημένους μας να ανέβουν εδώ στο βήμα και εγώ θα πω δύο λόγια για το ποιοι είναι αυτοί. Okay, so we're going to Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο κομμάτι αυτής της ακρόασης δίνοντας τον λόγο στον κύριο Μάρκος Χάρτμαν που είναι εισαγγελέα και επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης κυβερνοεγκλήματος στην Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, στην Κολονία. Έχουμε μαζί μας επίσης τον κύριο Πέτερ Σνάιντερχαν από την Γερμανική Ομοσπονδία Δικαστών και τον Γιάν Κέρχοφς από την Γενική Εισαγγελία του Βελγίου από τη Μονάδα Αντιτρομοκρατίας. Σας καλωσορίζω όλους. Και έχουμε και τον κύριο Μίτσελ μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε έτοιμες τις ε, διαφάνειες Κοντεύουμε όλοι να κοιμηθούμε, είναι 3 και 20. Λοιπόν, έχουμε τον Μάρκους Χάρτον μαζί μας. Όπως είπα, είναι εισαγγελέα και επικεφαλή της μονάδας καταπολέμησης, του κυβερνοεγκλήματο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία της Γερμανίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι. Θέλω να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική αναγκαιότητα που ε, συνδέονται με τις αναγκαιότητες που συνδέονται με το θέμα που συζητάμε σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω καταρχάς με ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι το θέμα που συζητάτε σήμερα είναι ένα από τα πλέον επιτακτικά, αν όχι το πιο επιτακτικό ερώτημα που με απασχολεί όσον αφορά την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων και, τη διεθνή συνεργασία. Γι' αυτό και είναι μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία να σας δώσω κάποιες ε, πρακτικές πληροφορίες. Θεωρώ δε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το ζήτημα αυτό να ρυθμιστεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με ομοιόμορφο τρόπο. Το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι στον, στο κυβέρνο έγκλημα δεν υπάρχει πλέον καμία διαδικασία που να υπόκειται αποκλειστικά σε εθνική αρμοδιότητα στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Ξανακοίταξα σήμερα με αφορμή την σημερινή ακρόαση ε, όλο το σύστημα διαδικασιών και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε μία δικαστική διαδικασία που να μην έχει με την μία ή την άλλη μορφή τη διάσταση της ε, διαστηνοριακής ε, συνεργασίας με τις αρχές άλλων χωρών. Και για να μπορείτε να ταξινομήσετε αυτές τις εμπειρίες μας με τον σωστό τρόπο, να σας ε, δώσω κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες από την καθημερινή εργασία της μονάδας μου. Η μονάδα μου στη Βόρεια Ρινανία Ρινανία-Βεστφαλία είναι μια κεντρική μονάδα για ε, την καταπολέμηση της, ε, του κυβερνοεγκλήματος. Με δύο λόγια μπορεί κανείς να πει ότι με 21 εισαγγελείς είμαστε υπεύθυνοι ε, για το κυβερνοέγκλημα σε μια επικράτεια στην οποία κατοικούν 18 εκατομμύρια άνθρωποι και το 1 τρίτο των μεγαλύτερων 100 ε, γερμανικών επιχειρήσεων. Και οι διαδικασίες που παρακολουθούμε και ερευνούμε είναι αποκλειστικά διεθνείς. Θέλω να σας δώσω και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή η αναφορά από ένα διαδικτυακό ε, περιοδικό αφορά μια μεγάλη έρευνα και επιχείρησή μας για την καταπολέμηση, για την δίωξη ενός botnet, δηλαδή ενός δικτύου ε, υπολογιστών ζόμπι, ε, μέσω του οποίου εγκληματίες προβαίνουν σε εκβιασμούς κτλ. κτλ. Εδώ αναδεικνύεται η διεθνής διάσταση. Ένας Βρετανός πολίτης με έδρα την Κύπρο κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε ένα, σε ένα λιβεριανό δίκτυο και εξαιτία αυτής της διαδικασίας της επιχείρησής του, του εγκλήματος που διέπρατε, έπεσε το ίντερνετ για εκατοντάδες ε, χιλιάδες χρήστες στη Γερμανία. Από αυτό και μόνο το παράδειγμα αποδεικνύεται ότι αν δεν υπάρχει ένα λειτουργικό διεθνές σύστημα, ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν υπάρχει περίπτωση καμία δικαστική ή εισαγγελική αρχή να μπορέσει αποτελεσματικά και επιτυχώς να διεξαγάγει τις της. Τις της. Εμείς τα καταφέραμε σε αυτή την περίπτωση, σε συνεργασία με τους αλλοδαπούς συναδέλφους μας και θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με τους ε, παράγοντες που οδήγησαν στην επιτυχία μου. Ε, είναι πολύ βεβαίω αυτοί οι παράγοντε, αλλά θέλω να επισημάνω και να, να αναδείξω κάποιου συγκεκριμένου. Πρώτον, ταχύτητα. Η ποινική δίωξη έχει έναν διοικό χαρακτήρα στο διαδίκτυο. Είναι 0 ή 1. Αν ή μάλλον άπαξ και διαγραφούν τα στοιχεία μιας ε, αξιόπινης πράξης, οι δικαστικές αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πια. Έχουν δεμένα τα χέρια τους. Και εδώ δεν μιλάμε για ημέρες ή εβδομάδες που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά για ώρες. Η οργάνωση των δομών, αυτών που σας περιέγραψα, των εγκληματικών, ε, αλλάζουν με την ταχύτητα του φωτός πολλές φορές. Ε, γι' αυτό και ε, χρειάζεται κανείς να μπορεί μέσα σε δύο ώρες ή έχει στη διάθεσή του μόνο δύο ώρες για να μπορέσει να έχει κάποιες ελπίδες οι έρευνές του να στεφθούν με επιτυχία. Αν δεν τα καταφέρει κανείς αυτό εντός δύο ωρών, πρόοδο δεν υπάρχει περίπτωση να σημειώσει στην έρευνά του. Και γι' αυτό είναι ύψης της σημασίας να ε, εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ε, ποινικών μας διαδικασιών. Εδώ θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία. Στη μονάδα μου είναι αυτονόητο ότι είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, να ζητούμε και να παρέχουμε τη βοήθειά μας ε, σε άλλες ε, δικαστικές, διοκτικές αρχές ε, των άλλων κρατών μελών. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν αυτή εξασφαλίζεται μόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς νομικές βάσεις. Γι' αυτό και χρειάζεται να ρίξουμε μια ρεαλιστική ματιά στο ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη συνεργασίας που οδηγεί μόνο κάτω από τις ανάγκες στην εξέβρεση λύσεων. Το να υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός εργαλείων θα διευκόλυνε τις διοκτικές αρχές στο έργο τους. Σημαντικά. Γι' αυτό να ρίξουμε μια ματιά στο ποια είναι τα υπάρχοντα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Φυσικά, λοιπόν, έχουμε εργαλεία, όπως έχουμε τις κοινέ ομάδες ε, διερεύνησης. Έχουμε κόμβους ε, εισαγγελέων, δηλαδή μορφές συνεργασίας εισαγγελικών δικαστικών αρχών στον, ε, στην Ευρώπη. Έχουμε τις, ε, την, την Ευρωπαϊκή Εντολή Ερεύνης. Όμως, αυτά τα κλασικά παραδοσιακά εργαλεία πρώτον χαρακτηρίζονται από αρκετά γραφειοκρατικό, από γραφειοκρατική φάση, φύση, είναι δυσκίνητες, ωστόσο από την άλλη πλευρά ε, υπάρχει ανάγκη να έχουμε γρήγορη πρόσβαση ε, στο διεθνές πλαίσιο, στο διεθνές διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο να σας πω και κάτι ακόμη για το ισχύο νομικό πλαίσιο. Φυσικά υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα σε εμά και τους διάφορους τηλεπικοινωνικούς παρόχους. Και βεβαίω είναι σημαντικό οι αρχές να μπορούν να διατηρούν αυτές τις καλές επαφές. Ωστόσο, η συνεργασία αυτή, ιδίω όσον αφορά τους Αμερικανούς ε, παρόχου υπηρεσιών, η συνεργασία λοιπόν αυτή έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Και αυτή η εθελοντική αρχή, προαιρετική αρχή, ακόμη και αν η συνεργασία είναι καλή, οδηγεί στο ότι εμπορικοί πάροχοι υπηρεσιών πολλές φορές δεν ερευνούν ή δεν μπορούν να ερευνήσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους για να μπορούν να απαντούν σε εμάς ε, στο σωστό χρόνο έγκαιρα. Γι' αυτό και για εμάς ο προαιρετικός ε, χαρακτήρας ε, είναι παροχημένος. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η πρόταση που ε, συζητούμε σήμερα ε, απαντούν σε αυτές τις ανάγκες των διοκτικών και εισαγγελικών αρχών. Φυσικά, έχω παρακολουθήσει τα υπέρ και τα κατά που έχουν αναδειχθεί στη συζήτηση. Και φυσικά μπορεί κανείς να πει πολλά σχετικά με την αλληλεπίδραση των διαφόρων προτάσεων, των υπαρχόντων εργαλείων και καταλαβαίνω πολλά, πολλές από αυτές τις ανησυχίες όσον αφορά για παράδειγμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ορθώς συζητούνται αυτά. Ωστόσο πρέπει να δοθεί κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία της νομιμότητας. Και να αναδείξω ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένω δεν έχει φωτιστεί αρκετά. Θέλω λοιπόν να σας πω γιατί δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε προαιρετικές διαδικασίες. Στις ε, ποινικέ διαδικασίες στο κυβερνοέγκλημα υπάρχει πάντοτε μια αλυσίδα ε, βημάτων που ακολουθούμε, ηλεκτρονικών βημάτων. Ένας κρίκος να σπάσει σε αυτή την αλυσίδα δεν θα μπορέσετε να καταλήξετε πουθενά στην έρευνά σας. Οι έρευνες στο διαδίκτυο είναι σαν να ψάχνει κανείς βελόνα στο άχυρα. Μόνο αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνολική αλυσίδα, όλους τους κρίκους, της διάπραξης μιας αξιόπινης πράξης στο διαδίκτυο, θα μπορέσουμε να εξαρθρώσουμε την, ε, την πράξη αυτή και να την διώξουμε. Και θέλω να επισημάνω και ένα άλλο στοιχείο. Στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοκτικών αρχών με τα παραδοσιακά εργαλεία εξασφαλίζεται ότι ως διοκτικές αρχές ε, έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ, διασυνοριακή μεταξύ των αρχών ε, άλλων ε, κρατών μελών. Πολύ συχνά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Η βελτίωση λοιπόν αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών θα μπορούσε να είναι μια λύση που θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα συνολικά του συστήματος που έχουμε στη διάθεσή μας. Συνολικά, εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο όπου το ελληπές νομικό πλαίσιο και ο προαιρετικός χαρακτήρας δικαιολογούν τη δημιουργία ενός συστήματος που θα ενισχύει ε, περαιτέρω την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ε, συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών. Γι' αυτό, παρά τις αμφιβολίες και τις ανησυχίε που ενδεχομένως έχουν εκφραστεί, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Και θέλω να συνοψίσω τα λόγια μου με αυτό που λένε πολύ συχνά οι πληροφορικάροι. Πολύ συχνά ε, πρέπει κανείς στον προγραμματισμό να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, για μένα, η διαδικασία που έχει ξεκινήσει, μόνο σε ε, καλύτερα από ό,τι έχουμε σήμερα αποτελέσματα θα μας οδηγήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας ε, μετά την ε, ακρόαση αυτή. τι, τι πιστεύεις ότι θα πετύχουμε ως αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χάτσμαν. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Πίτερ Σνάιντεραν από τη Γερμανική Ένωση Δικαστών. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Η ανάλυση του κυρίου Χάρτμαν είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Χρειαζόμαστε νομική ρυθμίση για τις διασυνοριακές έρευνες και μάλιστα γρήγορα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο το νομικό εργαλείο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σωστό. Ήθελα να απαντήσω και την ερώτησή σας, ε, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος ε, για έρευνα ανταυτού. Αυτό θα έχει στην πράξη το πλεονέκτημα να μην υπάρχει ο κατακαιρματισμός που υπάρχει στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της ε, Βουδαπέστης. Τίφεται λοιπόν το ερώτημα του κατά πόσον τι χρόνο χρειάζονται τα δικαστήρια για να μπορούν να λάβουν αποφάσεις εδώ. Φυσικά είμαστε κατά των χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται στους δικαστές. Χρειάζονται το χρόνο που χρειάζονται για να λάβουν μια απόφαση. Αλλά φυσικά αν τα κράτη-μέλη έχει υποχρέωση να έχει κάποιον δικαστή ε, ανά πάσα στιγμή προκύπτουν αυτές οι υποχρεώσεις. Υπάρχει. Αυτή η εναλλακτική ενδεχομένω για τη χρήση του πλαισίου, του νομικού πλαισίου για το Ευρωπαϊκό Έντελμα Ερευνών. Τι γίνεται λοιπόν ε, τι θα γίνει στο μέλλον αν εκδίδεται εντολή υποβολή στοιχείων. Καταρχάς έχουμε τις ε, προϋποθέσεις για την εκκίνηση μιας δικαστικής αγωγή, μιας ε, διαδικασίας. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχουν ε, ρυθμίσεις και διατάξεις για την αρμοδιότητα για αξιόπινες πράξει. Άρα η εκκίνηση τέτοιων έναμων διαδικασιών ε, εναπόκειται στο κράτο μέλο. Το θέμα του αξιοπίνου για τρία χρόνια είναι και αυτό θέμα τον μέλλον και το θέμα της αναλογικότητας. Άρα τελικά όλα αυτά ελέγχονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και ο κανονισμός ε, δεν δίνει καμία ευρωπαϊκή διάταξη προς την κατεύθυνση αυτή. Θα έπρεπε στους εθνικούς ε, νομοθέτες, ούτε στα δικαστήρια για την κανονισμό. Συνεχίζουν λοιπόν τα δικαστήρια να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε εθνικό επίπεδο και αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί ένα βασικό μειονέκτημα, ένα βασικό αδύναμο σημείο του κανονισμού, ένα από τα βασικά προβλήματα που θα δυσκολέψει όλους όσοι θα εργαστούν στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Έχω την εντύπωση είναι πολύ διαφορετικές και κατακριματισμένες οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις υποβολής τέτοιων, τέτοιες εντολής. Όταν λάβει κανείς λοιπόν μια εντολή υποβολή στοιχείων, πρέπει να ελέγξει κατά πόσον υπάρχει ε, προφανής ε, παραβίαση των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Τέτοιος έλεγχος είναι δυνατόν να γίνει αν ε, τα δικαστήρια του κράτους μέλους υποβολής ε, των, της εντολής ήταν, δεν έδειξαν τη σωστή προσοχή. Δεν ξέρω αν οι νομικές υπηρεσίες ε, των παρόχων μπορούν να έχουν την ε, δυνατότητα να κάνουν μια τέτοια, ένα τέτοιο νομικό έλεγχο, να λαμβάνουν τον ευθύνη καν. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι τύφεται το θέμα των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου που διακυβεύονται. Το πρόβλημα είναι, και αυτό είναι ένα σημείο κριτικής, το πρόβλημα είναι ότι η εφαρμοσιμότητα τέτοιων ε, εντολών τίθεται ένα σε αμφιβολία. Γιατί ο κατηγορούμενος μπορεί να υποβάλει δικαστικό αίτημα για την νομιμότητα της εντολής και ο εισαγγελέα είμαι εντελώ αντίθετα. Αντίθετο να υπάρχει ένα νομικό εργαλείο για την εκτελεσιμότητα του οποίου δεν ευθύνομαι εγώ δεν είναι δυνατόν να κάνω διάλογο με τον πάροχο για το κατά πόσον θέλει ή δεν θέλει να προβεί σε εκτέλεση της εντολής. Ο πάροχος θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει την να απαντήσει στο αίτημα. Το ότι υπάρχουν τεχνικές, ε, τεχνικοί περιορισμοί ε, είναι δεδομένο, αλλά δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε και για την νομιμότητα της εντολής. Άρα το βασικό, η βασική αδυναμία του όλου κανονισμού δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο πάροχος είναι υπεύθυνο ουσιαστικά για την σεβασμό των ασφαλών δικαιωμάτων του κατηγορούμενου, αλλά ότι δεν εγγυόμαστε την εκτελεσιμότητα της εντολής. Και κάποιες φορές μου θυμίζει το καθεστώς ε, νομικής αρρωγής, όπου είναι εθελούσιος ο χαρακτήρας. Άρα εδώ ουσιαστικά ο πάροχος μπορεί να ε, ισχυριστεί ανα πάσα στιγμή ότι δεν γίνονται σεβαστές οι διτάξεις των θεμελιδών δικαιωμάτων και ότι επιτεύχεται ένα αμφιβόλου νομιμότητα. Βάσει ποιων δικαιωμάτων πρέπει να ελέγξει τι τι θα πρέπει να διευκρινιστεί, με ποιο αποτέλεσμα, ποια δικαιώματα ελέγχονται σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο, τον πάροχο, το κάτω μέλος. Όλα αυτά δεν τα ρυθμίζει ο κανονισμός. Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να πρόκειται για ένα απόρριτο τέτοιο μέτρο, γιατί από τη στιγμή που ενημερωθεί ο κατηγορούμενος, φυσικά πάθουν να ισχύουν διάφορες συντάξεις. Αλλά φυσικά όσο με το γνωρίζει αυτό, ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να καταγγείλει την μη τήρηση ενδεχομένω των δικαιωμάτων του. Εδώ και πάλι ο κανονισμός δεν προβλέπει τίποτα. Υπάρχει ένα ένομο μέσο στο άρθρο 17 στα πλαίσια του παρόχου. Είναι ενδιαφέρον από πλευράς ένομων μέσων. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτό το ένομο μέσο μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί τα δεδομένα όταν εκδίδονται στην διαδικασία των ερευνών, αν αξιολογηθούν και στην πορεία προκύψει αφού ο κατηγορούμενος ε, γνωρίζει πλέον ότι έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα του αυτά, το θέμα είναι πώς ε, μπορούμε να επαναρθώσουμε, πώς μπορούμε να διαγράψουμε αυτά τα παρανόμως ε, συλλέχτα δεδομένα. Και εδώ σιωπή ο κανονισμός. Στο άρθρο 14, σχέση με τις τρίτες χώρες. Εδώ η δικαιοσύνη ε, το δικαστικό σώμα, πολύ απλά του δίδεται μια αρμοδιότητα την οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει. Η κλασική νομική αρρωγή να φροντίσει ότι οι πάροχοι θα ανταποκριθούν στις υποχρέωσεις, αλλά δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα του δικαστικού σώματος να διαπιστώσουν κατά πόσον η άρνηση χορήγηση των στοιχείων αυτών ναι, με σύμφωνα με το νομικό σύστημα μιας άλλης χώρας. Αυτό θεωρώ ότι επιβαρύνει υπερβολικά. Άρα έχουμε ερωτηματικά, σειρά ερωτηματικών, τα οποία προκύπτουν από τον κανονισμό. θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να συνδέονται με τη χώρα κατοικίας του κατηγορουμένου. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτό δεν μπορεί να το πετύχουμε σε ένα σύστημα μέσα στο Ευρωπαϊκό δέλεμα Ερευνών, προκειμένου να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε στα ερωτηματικά και στα κενά που έχει ο κανονισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πολύ κεντρικό, υπερβολικά κεντρικό ρόλο, τον οποίο έχει ο πάροχο, που δεν μπορεί να διαμορφωθούν τον τρόπο που προτείνει ο κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Συνάντραχαν, και νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει για του δύο πρώτου ομιλητέ, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτά. Και βλέπω ότι ο επόμενο ομιλητή μα είναι πολύ νευρικό. Θέλει και αυτό να πάρει το λόγο για να παρουσιάσει τη δική του άποψη. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον Γιάννη Κέρκοφ, δικαστή σε ομοσπονδιακό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο, σε Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελία. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ε, η εισήγησή μου, αν τα διαφάνεια μου έχουν ε, μπει εδώ, να υπάρχει μια παρουσίαση του κ. Κέρχου συνέτοιμη. Σας ευχαριστώ. Όπως ε, σωστά παρατηρήσατε κυρία Πρόεδρε, ανυπομονούσα να μπω και εγώ στη συζήτηση, διότι το θέμα ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, επειδή είμαι ομοσπονδιακός εισαγγελέα, το Γενικό Γραφείο του Βέλγου Εισαγγελέα. Καθημερινά ασχολούμαι με υποθέσεις ε, αντιτρομοκρατίας και κυβερνοεγκλήματος σε αρκετά μεγάλη κλίμακα. Επόμενη διαφάνεια. Στις 17 Απριλίου 2018 ήμουν ε, αρκετά ευτυχής διότι προσθέθηκαν νέα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας, προτάθηκαν μάλλον νέα εργαλεία που μου έδωσαν την αίσθηση πως μπορούμε και ότι έπρεπε να είχαν γίνει αυτά εδώ και καιρό. Αγνοήστε την ε, σημαία παρακαλώ σε αυτή εδώ τη διαφάνεια. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι η πρώτη που θα φυτέψει η σημαία στο νέφος και όχι στο φεγγάρι. Είμαστε ευτυχείς γιατί οι προτάσεις αυτές πράγματι ανταποκρίνονται στην ζήτηση. Θέλαμε να έχουμε συγκεκριμένα μέσα για να μπορούμε να συλλέγουμε στοιχεία τα οποία είναι τόσο εύκολο να διαγραφούν, να εξαφανιστούν. Πρέπει, όπως έλεγε η συνάδελφος, να δρούμε πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις αποδείξεις, τα αποδεικτικά στοιχεία και ανησυχούμε για τις ασφαλιστικές δικλίδες, τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής. Εγώ μάλιστα έχω πάρει όρκο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής Καθημερινά το προσπαθώ. Θεωρώ πως είμαι σαν ένας χειρούργος που κάποιες φορές για να θεραπεύσει πρέπει να κόψει. Θα πρέπει ωστόσο να έχω τον ιστέρι μου, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι καλή η εγχείρηση. Πρέπει ωστόσο κάπως να προσγειωνόμαστε από καιρό εις γιατί έχω την εντύπωση πολλές φορές ότι αυτή η ατμόσφαιρα δίνει την εντύπωση ότι ο κόσμος πρέπει να προστατεύεται από ανθρώπους σαν και εμένα. Μα δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι ισχύει όντω, ότι δηλαδή θα πρέπει όλοι να ε, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί παροχοί ε, υπηρεσιών στο ίντερνετ με όγκους στοιχείων για τα οποία ποτέ δεν θα είχαμε αρκετό ε, χαρτί για να γράψουμε για όλα αυτά. Ο κόσμος δίνει τα στοιχεία σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες από μόνος του και θα πρέπει να πάρα πολύ καλά να έχουμε υπόψη μας πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και δεν θεωρώ πως η λύση είναι να επιτρέψουμε στη ΣΥΠΑ να εισχωρήσουν στις δικές μας ερευνητικές ομάδες. Μάλιστα, με αυτήν εδώ την πρόταση θεωρώ πως θα μπορούσαμε κάποιους από αυτούς τους παίκτες να τους αναγκάσουμε να ε, συμμορφωθούν προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων και διάφορες ε, προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε εδώ στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ιδιωτική ζωή δεν είναι πάντοτε μέρημνα όλων. Είναι δική μου μέρημνα, δική σας μέρημνα, αλλά είναι και ένα προϊόν η ιδιωτικότητα. Εάν είστε ευχαριστημένος που πρέπει, δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να χρησιμοποιείτε το Google, αυτό είναι επειδή ε, παίρνουν τα στοιχεία σας. Ε, πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε να υπάρχουν ναι μεν ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά να μην θεωρούμε πως σε αυτή ε, την ε, ε, σκηνή του εγκλήματος, γιατί πρόκειται για μια γιγαντιά σκηνή εγκλήματος, να μην μας αφαιρείται τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κυνηγήσουμε τον κόσμο που κάνει αδικήματα στο ίντερνετ. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ζητήσουμε στοιχεία από αυτές τις εταιρείες, να απαιτήσουμε στοιχεία, γιατί είναι χώρος εγκλήματος, σκηνή εγκλήματος, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε τον ε, κύριο ηλεκτρονική ε, απόδειξη, μετά έχουμε την κυρία επιβολή του νόμου που κατά κάποιο τρόπο μένει εκτός της κατάστασης και δεν θέλω να ακουστώ από, ε, ως απεγνωσμένος, αλλά από τη μια πλευρά έχουμε την ταχύτητα της επικοινωνίας στο ίντερνετ, την πτυτικότητα των δεδομένων και της επικοινωνίας και από την άλλη έχουμε αδυναμία επιβολής του νόμου ε, έγκαιρα, αρκετά έγκαιρα ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Ευρωπαϊκό ένταλμα υποβολή στοιχείων. Αυτή είναι μια εικόνα με τους φακέλους μου στο γραφείο μου. Και θα ήθελα να καλέσω όποιον θέλει να έρθει να με επισκεφθεί, να διαλέξει έναν φάκελο και να προσπαθήσει να ανακαλύψει το φάκελο όπου δεν χρειαστήκαμε δεδομένα. Και μάλιστα ε, πρόσβαση στα δεδομένα και πολύ γρήγορα. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε την πρόταση. Άμεση συνεργασία ανάμεσα στα ε, Υπουργεία Δικαιοσύνης, τις εγγελίες και τους παρόχους ε, ε, υπηρεσιών ίντερνετ. Όμως εκπρόσωπος στις, στην Ένωση έχουμε το ε, την έδρα των περισσότερων εταιριών στις ΙΠΑ. Ε, η μία απάντηση δίνεται σε 10 μέρες, αλλά σε 6 ώρες όταν είναι επίγουσα η περίσταση. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την ευκαιρία που ε, έχουμε να ζητήσουμε στοιχεία άμεσα προς τις παρόχους και αυτή είναι τη θέμενη αξία του συγκεκριμένου μέσου. Πρόκειται για νέα ιδέα. Διότι νωρίτερα στην αρχή αυτής της συνεδρίασης ε, προτάθηκε πως αυτή η ιδέα είναι τελείως νέα, αλλά δεν είναι. Είναι νέα για την πρόσβαση στα δεδομένα, είναι νέα όσον αφορά τα δεδομένα για τις συναλλαγές, αλλά για τις βασικές πληροφορίες του συνδρομητή από το 2001 με το άρθρο 18.1β τη Σύμβασης της Βουδαπέστης έχουμε τις βασικές πληροφορίες του συνδρομητή και ισχύει η ίδια αρχή. Πρόκειται για 17 χρόνια τώρα που λειτουργεί αυτή η ε, αρχή. Έχουμε νομίζω 60 χώρες που έχουν κυρώσει την σύμβαση της Βουδαπέστης. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα με βάση τη σύμβαση να μπορεί κανείς να ανακτήσει τις βασικές πληροφορίες για το συνδρομητή άμεσα από τον πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ σε άλλη χώρα. Η πρόταση λοιπόν που είναι επιτάπητος απλώς προχωρά περισσότερο όσον αφορά την αρχή που ήδη εφαρμόζεται ε, εδώ και 17 χρόνια. Πρέπει να το γνωρίζουμε λοιπόν ότι εάν και κατά κάποιο τρόπο κάνουμε διαφορετική εξολόγηση για το τι θα πρέπει να κάνουμε με την αρχή της άμεσης πρόσβασης ε, ε, σε στοιχεία ενός παρόχου υπηρεσιών ίντερνετ σε μια άλλη χώρα, να γνωρίζουμε πως αυτή την αρχή ήδη την έχουμε εγκρίνει στη Σύμβαση της Βουδαπέστης πριν 17 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τις ε, σχέσεις του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Έρευνας ε, έναντι του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Υποβολής Στοιχείων, όταν κανείς κάνει εγχείρηση ματιού, ρωτάει, προτιμάτε να χρησιμοποιήσουμε το ψαλίδι, το νηστέρι ή το λέιζερ. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα μπορούσαμε με το ψαλίδι να το κάνουμε, αλλά δεν θα ήταν κατάλληλο και μάλλον δεν θα έχει ωραία όψη, αλλά ούτε θα είναι αποτελεσματική εγχείρηση. Χρειάζεται, συμφωνώ απολύτως, με τον συνάδελφο Χάρτμαν, που εστίασε στην ανάγκη του συγκεκριμένου μέσου, και θα σας δώσω πολύ συγκεκριμένα και σαφή παραδείγματα. Εδώ έχουμε ε, περιπτωσιολογικά παραδείγματα τρομοκρατίας όπου προσπαθούσαμε να προλάβουμε μία τρομοκρατική επίθεση στη βιολογική, σε βιολογικό έδαφος. Εκεί ζητήσαμε από την ε, Ανακριτική Επιτροπή στις ΙΠΑ Πήγαμε δηλαδή στις ΙΠΑ στις 7 Οκτωβρίου 2016. Ανακαλύψαμε στην εκτέλεση της Ερευνητικής Επιτροπής ότι ένας από τους υψηλά ιστάμενους αξιωματικούς ε, στο Ισλαμικό κράτος χρησιμοποιούσε συγκεκριμένο λογαριασμό hotmail για να στέλνει τις εντολές του και βεβαίως αυτό ε, ε μας... Ε, προκάλεσε την προσοχή. Τι κάναμε, παγώσαμε γρήγορα το συγκεκριμένο λογαριασμό. Προτείναμε δηλαδή Microsoft να, να παγώσει όλα τα πάντα γύρω από αυτόν τον λογαριασμό Hotmail. Ο, θεωρήσαμε πως όλοι θα ήταν υπέρ του να παρεμποδιστεί μια τρομοκρατική επίθεση. Η, το αίτημα έμλατ υπευλήθη τον Οκτώβριο του 2016 στη ΣΥΠΑ. Περιμέναμε και ζητήσαμε, ρωτήσαμε το Υπουργείο Δικαιοσύνη, τον είπα πώ πάει, έχουμε νέα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνη τη ΕΠΑ είναι πολύ πρόθυμο, αλλά και εκεί έχουν ε, μεγάλη συμφόρηση γιατί όλοι οι μεγάλοι πάροχοι βρίσκονται εκεί, έχουν παγκόσμιους παίκτες στην επικράτειά τους, πρέπει να καταθέσουν εντάλματα στα τα οποία εγκρίνονται από το δικαστήριο. Έγινε λοιπόν συζήτηση και έπειτα ένας δικαστής της ε, ενέκρινε την παράδοση των συντηρημένων διατηρημένων στοιχείων και λάβαμε τα αποτελέσματά μας στις 7 Νοεμβρίου του 2017. 12 μήνες και 26 μέρες αργότερα. Και δεν είναι αυτό η εξαίρεση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στις 7 Νοεμβρίου 2017 μας είπαν ότι αυτός ο λογαριασμός είχε ήδη διαγραφεί στις 26 Μαΐου του 2016, πριν δηλαδή και από την εντολή διατήρησης. Οπότε σε εκείνη την φάση καταλαβαίνετε ότι έχεις βλεχτεί μέσα σε ένα σύστημα που δεν ξέρεις καν τι ίδιους στοιχεία να περιμένεις και πρέπει να περιμένεις πάρα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα για να πάρεις απαντήσεις. Και μετά ρωτάει κανείς, πώς το λύνεις αυτό με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Ερεύνης ή την αμοιβαία νομική συνδρομή. Και μου άρεσε η ερώτηση που έθεσε η κυρία Ιντεφελτ νωρίτερα στον καθηγητή Μπέζε. όπου αφορούσε τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και τότε θα πρέπει να προτείνουμε μια λύση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και υπόθηκε ότι ναι, έχουμε λύση και έχουμε το MLA και έτσι λειτουργεί το MLA. Ναι, αυτό για περιπτώσεις τρομοκρατίας και για περιπτώσεις όπου έχουμε ανθρώπους που έχουν συλληφθεί και περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτές είναι μια πραγματικές διαδικασίες Δεν λειτουργεί όμως πραγματικά. Υπάρχει λύση και η λύση είναι η συζήτηση επιτάπητος. Ναι, ναι, θα κλείσω, θα κλείσω. Υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Έτοιμα διατήρησης Ισπανίας προς το Βέλγιο στις 17 Δευτέρου 18 για βασικές πληροφορίες συνδρομητή και δεδομένα πρόσβασης για τους τελευταίους 9 μήνες. Έχουμε ε, ένταλμα που εκδόθηκε το Μάρτιο, υποβλήθηκε στο Βέλγο δικαστή και πάει πίσω εννέα μήνες. Όμως οι Νέα μήνες λόγω της, ε, των περιορισμών ε, παρακράτησης στοιχείων στο Βέλγιο 15 Απριλίου μπορεί να πάει πίσω εννέα μήνες και όχι από την ημερομηνία διατήρηση. Οπότε ήδη εδώ υπάρχει πρόβλημα και όταν εκτελείται στα τέλη του Μαΐου Υπάρχει το πρόβλημα ότι εντωμεταξύ ο λογαριασμός μπορεί να έχει διαγραφεί και ούτως ή άλλως την εκτέλεση. Τη εντολή έρευνη θα είσαι πίσω. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις κάθε μέρα έτοιμα διατήρησης και την καλύπτεις όλες τις μέρες μέχρι το τέλος. Είναι αυτό λύση όμως δεν νομίζω πως είναι πραγματικά λύση που να είναι αποδεκτή. Και έπειτα και το πρόβλημα της κοινοποίηση. Πολλοί θεωρούν ε, ότι πρέπει να υπάρχει η κοινοποίηση, όμως ε, στην πράξη να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι θα συμβεί. Η Ρουμανία κάνει ένα αίτημα ε, υποβολή στοιχείων στην Microsoft που έχει έδρα στο Βέλγιο. Η Ρουμανία λέει πως δεν υπήρχε στόχος ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο ύποπτος. Οπότε πρέπει να κοινοποιήσουμε το, την χώρα επιβολής του νόμου. Άρα γίνεται μια κοινοποίηση. Και τι θα γινόταν αν άρχιζε όλη η Ευρώπη να κοινοποιεί το περιεχόμενο των ετοιμάτων της προς τη Microsoft και προς το Βέλγιο. Ο ύποπτο που είναι στη Γαλλία θα σκάσει τα γέλια. Αυτό θα συμβεί. Θα έχουμε ένα βουνό κοινοποίηση. Το θέμα λοιπόν είναι τι θα κάνουμε όλες αυτές τις κοινοποίησεις. και δεν έχουμε καμία ταυτότητα για το ποιο είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν έχουμε ιδέα. Ναι, 50 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Άρα λοιπόν τις περισσότερες φορές χρειαζόμαστε απλώς τα δεδομένα για να γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Εάν λοιπόν φτιάξουμε κανόνες που εμείς πρέπει να το θέσουμε στην πράξη σε λειτουργία, το πού θα είναι ο άνθρωπος δεν θα είναι τόσο εύκολο να βρεθεί. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε με το βουνό των κοινοποιήσεων χωρίς νόημα. Δεν ξέρω. Είναι ένα μεγάλο βουνό, ένα μεγάλο σφόρτος εργασίας, γιατί αποφασίσαμε να μην εμπιστευτούμε τον συνάδελφο από τη Ρουμανία. Είναι λοιπόν αυτό ζήτημα. Και η τελευταία μου διαφάνεια. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, θα είμαι λίγο δυσάρεστη με κάποιους συναδέλφους, αλλά μας τελειώνει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Τουλάχιστον ε, αν κάτι κρατάμε είναι ότι δραστηριοποιήσετε ενεργά στον τομέα αυτό. Για άλλα ε, στοιχεία της παρουσίασής σας δεν, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησαν τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση ε, καλό είναι να προσφέρει ο καθένας τη δική του οπτική στη συζήτηση. Θέλω να γίνει συζήτηση με τους συναδέλφους ευρωβουλευτές, αλλά έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ιαν Μίτσελ, που είναι ε, πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ακούσουμε και την δική του παρουσίαση και μετά θα προχωρήσουμε σε ερώτα απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε εξαιρετικές εποχές ε, απαιτούνται εξαιρετικά μέτρα. Ε, και αυτή η ρίση πάντοτε ε, ε, ίσχυε στον ιστορικό, στην ιστορία του ανθρώπου. Το ίδιο ίσχυε ακόμη και στην, στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η οποία ήταν, όπου η Γερουσία ήταν εκείνος ο οποίος εξέλεξε τον δικτάτορά της, τον πρώτο, όταν και ο όρος αυτός σήμαινε απλώς έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύεσαι. Ακούσαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση από τον κύριο Κέρχοφ και από τον κύριο Χάρτμαν ότι ζούμε σε ε, ε, εξαιρετικές εποχές ε, και γι' αυτό χρειάζονται εξαιρετικά μέτρα. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και πιο νόμιμα και αναλογικά μέτρα για να επιτύχουμε τον ίδιο στόχο. Και αυτό κρύβεται και πίσω από τις προτάσεις της CCBE του Συμβουλίου των Διοικητικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ε, μακροσκελές έγγραφο το οποίο έχετε όλοι λάβει, αιτιολογημένο και ε, βεβαίω σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σα το παρουσιάσω με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω είναι ποια είναι τα βασικά προβλήματα που εντοπίζουμε εμείς στην ε, πρόταση της Κομισιόν και που μας οδηγούν ε, στο να έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι η απάντηση που δίνεται στο πρόβλημα δεν είναι αναλογική. Πρώτον, Υποτίθεται ότι η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν το άρθρο αυτό είναι η σωστή νομική ε, βάση διότι ε, δεν εξασφαλίζει την συνεργασία μεταξύ των νομικών συστημάτων. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τη δομή, την αρχιτεκτονική των προτάσεων. Διότι επί της ουσίας αυτό που έχουμε είναι ότι το κράτος έκδοσης μπορεί να εκδίδει την εντολή του ε, στο επίπεδο της δικαστικής εξουσίας, αλλά μπορεί και όχι. Απευθύνει λοιπόν όχι, την εντολή του όχι σε κράτος εκτέλεσης, αλλά σε ιδιώτη, σε ένα πάροχο υπηρεσιών. Έχεις λοιπόν μια, ένα διασυνοριακό αποτέλεσμα, το οποίο ε, δεν έχει προηγούμενο. Άκουσα ότι έγινε αναφορά στην ε, σύμβαση της ε, Βουδαπέστης, όμως αφορά μόνο τα δεδομένα ε, συνδρομητών, όχι τα δεδομένα περιεχομένου. Γι' αυτό πρέπει κανείς να έχει υπόψη το αυτή τη λεπτή διάκριση. Το βασικό πρόβλημα με την αρχιτεκτονική που σας παρουσίασα είναι ότι δεν υπάρχουν δικαστικά μέσα ελέγχου ε, στην ε, χώρα εκτέλεσης. Και στην πρόταση δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέεται με τα δεδομένα συνδρομητή και τα δεδομένα πρόσβασης. Θεωρώ ότι δεν συνάδει η πρόταση αυτή με τις υποθέσεις Benedict εναντίον Σλοβακίας και άλλες ε, υποθέσεις αποφάσεις του δικαστηρίου όπου επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης. Μπορεί κανείς να συγκρίνει και τα κείμενα της αρχικής πρώτης κομισιόν και της, της αναθεώρησης που έκανε το Συμβούλιο. Το αρχικό κείμενο της κομισιόν ήταν αρκετά κακό το οποίο κατάφερε και επιδίνωσε έτσι περαιτέρω η πρόταση της Προεδρίας του Συμβουλίου. Εξετάζουμε λοιπόν ε, το εξής. Ο παραλήπτης της εντολής, ο πάροχος εν προκειμένου, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό το έδειξε και η προτελευταία προ, διαφάνεια του ε, τελευταίο ομιλητή ε, για τη Microsoft, που είναι και ο λιγότερο ανησυχητικός πάροχος. Δεν έχουν καμία ιδέα οι πάροχοι αν συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες τους, οι οποίες τους ζητούνται παραβιάζουν θεμελιωδή δικαιώματα υπό το άρθρο 8 ή υπό το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, τα οποία και έχουν απόλυτο χαρακτήρα το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και, το, και την αποκλειστική προστασία που παρέχει το άρθρο 6. Δεν υπάρχει καμία εξορροπητική διαδικασία που να προβλέπεται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο πάροχος δεν έχει καμία, δεν έχει καμία δυνατότητα να σχηματίσει μία ε, συγκεκριμένη εικόνα, γνώμη. Ούτε και το ε, κράτος έκδοσης. Ενώ λοιπόν στην αρχική πρόταση υπάρχει δυνατότητα προσφυγής, όταν η εντολή αυτή παραβιάζει τον, τον χάρη θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπάρχει πλέον ένα πρόβλημα στο κείμενο της Προεδρίας. Και υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Ότι η αρχική θέση στο κείμενο της, της ε, Κομισιόν είναι ότι ο πάροχος έχει την ελευθερία να πει στον πελάτη του ότι έχει παραδώσει τα στοιχεία του εκτός αν λάβει οδηγίες περί, του αντιθέτου. Όμως, στην αφιερωμένη εκδοχή του κειμένου από πλευράς Προεδρίας η δυνατότητα του παρόχου διαγράφεται πλήρως. Και το σκεπτικό είναι ότι άπαξ και γίνει ε, μια, ε, ένα αίτημα, πρέπει και να εκτελείται. Και τέλος, αυτό ε, δεν θα το χαρακτηρίζα και εξισορρόπηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, η βασική θέση είναι ότι δεν ενημερώνει τον πελάτη. Εμείς θα λέγαμε επί της ουσίας ότι αν ε, είναι να θεσπιστεί κάτι τέτοιο, έστω και με ε, αμφισβητούμενη νομική βάση, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον απέτηση το κράτος μέλος έκδοσης μέσω, μέσω ε, δικαστικής προσφυγής να εξασφαλίζει και να αιτιολογεί για ποιο λόγο οι ε, πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν ε, κρυφές, εμπιστευτικές για λόγους ε, ε, που σχετίζονται με την έρευνα. Υπάρχουν και κάποια πρακτικά θέματα για το πώς θα παράγονται τα δεδομένα αυτά, αν θα είναι μηχανικά δεδομένα, πώς θα υποβάλλονται. Δεν υπάρχει ούτε καν επαρκής ορισμός των αποδεικτικών στοιχείων. Θα μπορούσαν να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία ε, κάθε είδους στοιχεία, ηλεκτρονικά και μη. Αυτά επίσης πρέπει να τα συζητήσουμε ε, περισσότερο. Νομίζουμε ότι δεν είναι καθόλου αναλογικές αυτές οι διατάξεις που προτείνονται. Επίσης, το έγγραφο της Προεδρίας, το οποίο χαιρετίζουμε βέβαια, έχει ένα στοιχείο, το συγκεκριμένο στοιχείο που χαιρετίζουμε, ότι ε, δεν υπάρχει κατάλογος του τι αποτελεί σοβαρό ε, έγκλημα. Αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, επίσης ούτε εδώ λύνεται το θέμα της πρόσβασης σε δεδομένα περιεχομένου. Και επίσης δεν υπάρχει και κάποιος ανασταλτικός μηχανισμός ε, ή ένας ε, μηχανισμός ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας. Ε, περιγράφεται το πώς εκδίδεται μια τέτοια εντολή, αλλά δεν περιγράφεται το πώς θα ολοκληρώνεται η πορεία της. Να σας πω εντάχει Πώς μπορούμε να τετραγωνίσουμε, τετραγωνίσουμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο με αναλογικό τρόπο. Υπήρξε μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να θεσπιστεί κανονισμό ή οδηγία. Το άρθρο 82 δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για την έκδοση, για την θέσπιση ε, κανονισμού ή οδηγίε. Ίσως αυτό είναι ίσονο ε, σημασίας. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα όσον αφορά τη χρήση του 82.1 ω νομική βάση. Όμως, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ε, επίγουσες περιπτώσεις όπου πρέπει να λαμβάνονται δεδομένα μέσω εντολής διατήρησης αρχείων, θα μπορούσαμε να δεχτούμε τη συγκεκριμένη πρόταση με κάποια εχέγγυα. Το επόμενο, το επόμενο στάδιο όμως για μας είναι προβληματικό γιατί φαίνεται ότι η εντολή υποβολή στοιχείων δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις ε, αρχές της ε, επικουρικότητας και με τα εθνικά νομικά συστήματα. Ως CCB θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, χρήση των EMLAT. Ξέρω ότι ακούστηκε εδώ στη συζήτηση, αλλά εδώ μιλούμε για τις ενδοευρωπαϊκές υποθέσεις, όχι για τις διασυνοριακές και ιδίως εκείνες με τις ΕΠΑ. Μπορούν λοιπόν να βελτιωθούν οι EMLAT μέσω ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της θέσπισης ταχύτερων διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, ε, το Ευρωπαϊκό Έντελμα Έρευνας είναι ένα θετικό εργαλείο, διότι η εντολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, πρότυπο για να ε, διερευνώνται εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις όπου ε, υπάρχουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Θεωρούμε ότι το εργαλείο αυτό είναι πολύ καλύτερα ισορροπημένο, έχει, συνοδεύεται από πολύ καλύτερα έχει Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι ε, οι εξαιρετικές εποχές δεν απαιτούν απαραίτητο εξαιρετικά μέτρα. Απαιτούν μέτρα τα οποία θα είναι αναλογικά και που θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές του κράτους δικαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Και θεωρούμε ως CCBE ότι όλοι οι στόχοι αυτοί μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς τη χρήση αυτών των νέων προτινόμενων εργαλείων. Ευχαριστούμε πολύ και όπως είπα και νωρίτερα έχω και εγώ αρκετές ερωτήσεις. Κανονικά ο πρόεδρος δίνει τον λόγο στον ε, εισηγητή, την εισηγήτρια. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή και προεδρεύω και είμαι εισηγήτρια θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα σε άλλους συναδέλφους μου. Η κυρία Ιντβελτ θέλει να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να απαντήσω καταρχά στην παρουσίαση του κυρίου Κέρκοφ. Κύριε Κέρκοφ, νομίζω ότι μα δώσατε όλα τα επιχειρήματα που χρειαζόμασταν για να καταψηφίσουμε την πρόταση αυτή. Δεν. πώ ξέρετε τι ταινίε με τον Τερτιχάρη. Εσεί κάπω προ τον φέρνετε. Έχετε τέτοια αποδεκτικά στοιχεία στα χέρια σα. τόσοι λίγη σεβασμό έχετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Είσαστε κίνδυνος για το κράτο δικαίου. Είσαστε καουμπόι. Και πραγματικά σοκάρομαι. Ήμουν λίγο λιγότερο σοκαρισμένη, λιγότερο, αλλά πολύ λίγο, από τις δηλώσεις του κ. Χάρτμαν. Όχι, όχι, ναι, επανέλθω στα δικά σχόλια. Είπατε ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να προστατεύονται από ανθρώπους σαν και εμένα. Προφανώς και χρειαζόμαστε προστασία. Δεν πιστεύω ότι οι λύσει στα πρόβληματα, τα οποία σωστά τα επισημάνατε, δεν πιστεύω ότι οι λύσει στα προβλήματα αυτά είναι να ξεπουλήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Εδώ μιλάμε για δικαιώματα. Δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτήσει οι Ευρωπαίοι πολίτε. Προφανώ δεν σα εντυπωσιάζουν από ό,τι βλέπω. Γιατί βλέπετε ότι είναι πολύ αργή η διαδικασία. Βάζω το ένα παράδειγμα ενός έτους και 26 ημερών που χρειάστηκε να περιμένετε. Αλλά δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν δύο πολύ Δεν θα φανταζόσασταν ότι δύο δημοκρατικέ χώρε στον κόσμο, πλούσιε χώρε, θα έπρεπε να σεβαστούν ένα τέτοιο, μια τέτοια προθεσμία. Κατά δεύτερον, Δεν είμαι ε, κατά του να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω ότι είστε συγκλονισμένο από αυτά που σα λέω, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει νομική προστασία για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και συνήθω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά προτείνει δημιουργία ειδικών αρμοδιοτήτων ε, για ανθρώπους ε, όπως εσείς και μετά για τους Ευρωπαίους πολίτες που δεν εφαρμόζονται τελικά. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα εφιστάμενα μέσα και μετά αν χρησιμοποιήσουμε και αν δημιουργήσουμε καινούργια μέσα θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη νομική προστασία για τους πολίτες. Γιατί όταν λέτε ότι είναι πολύ αργή η διαδικασία αυτή, πρέπει να μπούμε κατευθείαν στον τομέα του εγκλήματο. Κύριε Χάρτμαν, μιλήσατε μόνο για το έγκλημα. Η πρόταση όμω, δεν περιλαμβάνει μόνο το έγκλημα. περιλαμβάνει όλα τα είδη εγκλήματο. Και το επιχείρημα ότι όλα τα τεκμήρια μπορούν να εξαφανιστούν ε, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ισχύει, αλλά όχι για όλε τι περιπτώσει. Γιατί εγώ έχω υπόψη μου και άλλε περιπτώσει κυβερνήσει των κρατών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κυνηγούν με κοιό, που επικρίνουν την εκάστοτε κυβέρνηση ή κρατημέλη, όπου για παράδειγμα η άμβλωση αποτελεί έγκλημα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να διώξουν τι γυναίκε, για παράδειγμα, ή τα ισμικιό. Δεν ακούω τίποτε να μας λέτε για αυτά. Κύριε και λέτε και παραθέτω ότι το διαδίκτυο είναι μία τεράστια ε, σκηνή εγκλήματος. Μα τι λέτε, όλος ο κόσμος είναι μία σκηνή εγκλήματος. Υπήρχε και έγκλημα πριν από το ίντερνετ. Το φαντάζεστε. Ο κ. Σάντρεχαν μας ικανοποίησε με ευχαρίστησε με την ε, παρουσίασή του και γιατί ήταν πολύ πιο πολλές οι αποχρώσεις. Νομίζω ότι αν η Γερμανική Ένωση Δατικαστών είναι επικριτική για την πρόταση αυτή, θα πρέπει να δείξει προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ τεκμηριωμένες ανησυχίες και καλωσορίζω αυτά που είπε ο κ. Μίτσελ. Προφανώς ε, δεν υποβάλλατε εσείς την πρόταση, αλλά άτομα και εσάς θα κληθούν να την χρησιμοποιήσουν και μέχρι ότου βεβαιωθώ ότι δεν θα υπάρξουν καταχρήσεις, δεν πρόκειται να την υπερψηφίσω. Ευχαριστούμε, Σοφή. Και νομίζω ότι είναι πολύ και πολύ παθιασμένοι οι ομιλητές από διάφορες πλευρές. Ε, να έχετε υπόψη σας ότι πρόκειται για ακρόαση και ως εκ τούτου έχουμε προσκαλέσει διάφορους ομιλητές για να παρουσιάσουν ακριβώς αυτές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και να κάνουμε μια συζήτηση αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχουμε τρεις επιπλέον ομιλητές, η κυρία Ένστ, Μέλο και ο εισηγητή. Η Κορνιλία Ένστ έχει το λόγο. Οι πολλές όμορφες εικόνες είδαμε. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν μα βοηθάει φυσικά ιδιαίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω κάποιε ερωτήσει να κάνω. Καταρχά. το είπε και ο κ. Σνάιντερχαν ξεκάθαρα, υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικά νομικά συστήματα. Το κλασικό παράδειγμα, ένα αυστριακό λέει για παράδειγμα ότι δεν θέλει να εκδώσει ένα κατηγορούμενο γιατί δεν αποτελεί αυτό έγκλημα για την Αυστρία, ενώ για μα αποτελεί αυτό έγκλημα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά νομικά συστήματα. Πώ είναι δυνατόν ένα τέτοιο μηχανισμό να λειτουργήσει λοιπόν σε ό,τι αφορά διασυνοριακέ έρευνε. Και τώρα προ τον συνάδελφο, τον κύριο Χάρτμαν και τον κύριο Κέρκοφ, θα ήθελα να ρωτήσω πόσε τέτοιε περιπτώσει από αυτέ που παρουσιάσατε έχετε ζήσει, έχετε αντιμετωπίσει στη ζωή σα. Είναι η μοναδική περίπτωση αυτή, είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια παραπάνω από Τρίτη ερώτηση. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Χάν σε ό,τι αφορά τον εθελούσιο χαρακτήρα. Δεν υπάρχει εθελούσιο χαρακτήρα. Τι γίνεται αν ένα παρόχο πει όχι. Δεν μπορούμε μετά από έλεγχο τη σχετική νομική υπηρεσία διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να παρέχουμε τα στοιχεία αυτά. Τι θα σήμαινε αυτό, Πώ θα λειτουργούσε το σύστημα, Τελευταία ερώτηση και πάλι προ τον κύριο Χάν και τον κύριο Μίτσελ το Ευρωπαϊκό Τέλμα Ερευνών αναφερθήκε πολλά και είσαι. Τι θα αλλάζατε, όχι στον κανονισμό αυτό, αλλά τι θα αλλάζατε στο ένταλμα ερευνών. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη τροποποίηση σε ό,τι αφορά την πιο γρήγορη εκπαιδεύση. Ευχαριστούμε την ε, Κορνιλιά. Είναι στο κύριο Μέλλο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ και θα μιλήσω πορτογαλικά. Thank eh, e ευχαριστώ. Ακούγοντας τις εισηγήσει που κάνατε, πιστεύω πως το πρώτο δικαίωμα του πολίτη είναι το δικαίωμα να ζει σε ασφάλεια. Το δεύτερο είναι να γνωρίζει ότι οι εγκληματίες μπορούν να δικαστούν και να τιμωρηθούν όπου και αν βρίσκονται. Τρίτο δικαίωμα είναι το να γνωρίζει ότι οι πολιτικοί, οι βουλευτές, δεν δεσμεύονται περισσότερο για να υπερασπίσουν τις εγγυήσεις για τους εγκληματίες από ότι για τη δικαιοσύνη που θα πρέπει να ασκηθεί υπέρ του θύματος. Το έγκλημα δεν καταπολεμάται με τις κοινοβουλευτικές αγορεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε οι πρώτοι που θα εγγυηθούμε το σεβασμό για την εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών και με αποτελεσματικότητα να συλλαμβάνουμε και να κρίνουμε ε, τους εγκληματίες αλλά και να αποφεύγουμε τη διάπραξη νέων εγκλημάτων, σοβαρών εγκλημάτων. Αυτό δεν σημαίνει παραβίαση των ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σπάνια η κοινοβουλευτική αγόρευση ε, έχει προκαλέσει τόσο ζημιά όσο για εγκλήματα που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Πολλά λοιπόν από τα λόγια που λέγονται εδώ μέσα, για παράδειγμα για το PNR, την καταγραφή δηλαδή των ε, ονομάτων των ε, επιβατών των αεροπορικών ε, εταιριών, αυτοί που επίεζαν για να εγκριθεί αυτό το μέσο από το Ευρωκοινοβούλιο, με αυτά τα επιχειρήματα μας έψαν να το απορρίψουμε. Και ένας σοσιαλιστής, ο πρόεδρος της ε, Γαλλίας, μετά όμως από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που δέχτηκε η χώρα του, επέμεινε και απέτησε την έγκριση αυτού του PNR. Δεν ήταν ε, η μαγική σφαίρα του Ντέρτι Χάρη που καταπολέμησε το έγκλημα, αλλά η ανάγκη ε, που οδηγεί στο να κάνουμε ε, κάποιες αλλαγές. Εγώ σε, ε, σας λέω ότι ήμουν ανέκαθεν υπέρ του PNR. Ήμουν ανέκαθεν ε, υπέρ του PNR όταν άλλοι ε, μιλούσαν και βγάζαν λόγους επιλόγων υπέρ των ε, προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων. Ναι, αλλά κύριε Μέλο, μπορείτε να μας πείτε κάτι γνώμη σας για το σημερινό θέμα. Ναι, να σας πω... Όμως την προοπτική μου για να καταλάβετε γιατί υπολογίζω. Εντάξει, το PNR για μένα έχει σχέση, γιατί εγκρίθηκε τελικά. Και όπως σας είπα, ε, είχαν ακουστεί τότε τα ίδια επιχειρήματα. Πρέπει λοιπόν να έχει έχουμε εγγύηση ότι εκείνος που ερευνά τα εγκλήματα θα μπορεί να προστατεύσει εμένα και τους συμπολίτες μου. Μήπως θεωρείτε πιο αποτελεσματικό αντί για ένα νέο μέσο, αυτό το οποίο ε, συζητάμε εδώ, το, τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, μήπως ε, θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης να μπορεί να εκδοθεί με λιγότερα αίτια έκδοσης, γιατί εδώ μιλάμε για ιδιαιτερότητες των αποδεικτικών στοιχείων, μιλάμε για το ίντερνετ, μιλάμε για ε, ταχύτητα διερεύνησης και ε, κράτησης των στοιχείων, μήπως λοιπόν μέσω αυτής της του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Ερεύνης, λόγω αυτών των ε, ε, ιδιαιτεροτήτων θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτό το ένταλμα από μεθοδολογικής άποψης. Ε, αυτή είναι η ερώτησή μου. Μήπως λοιπόν θα ήταν πιο σκόπιμο το να αλλάξουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να καταλάβατε ε, αυτό το παράδειγμα που έφερα με το PNR, ότι δηλαδή η πολιτική πολλές φορές ε, μπορεί να καθυστερήσει τη λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μέλλο. και φυσικά αντιλαμβάνομαι και θυμάμαι πάρα πολύ καλά την Ευρωπαϊκή Οδηγία PNR. Την καταψήφισα και ακόμα πιστεύω και ακόμα επιμένω σε αυτή την απόφαση, αλλά προφανώς πάντα χρειάζεται να ελέγξουμε κατά πόσον χρειαζόμαστε νέα μέτρα ή να ενισχύσουμε ήδη φυστάμενα μέτρα. Είναι δύσκολο αυτό. Ο κ. Φραντς, ένας διαφορετικός ο ομιλητής. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Χάρτμαν. Είπατε ότι θέλετε να έχετε έναν ε, δικαστή για αιτήματα από άλλα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη συνεργασία αυτή. Μπορείτε να μας πείτε λίγο παραπάνω πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η συγκήτρια θα ήθελε και αυτή να πάρει το λόγο για να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κέρκοφ για το γεγονός ότι ανέφερε ότι θεωρούμε ότι η υπηρεσία της Facebook είναι δωρεάν. Και συμφωνώ, θα χρειαζόμασταν ρυθμίσει πολύ καιρό τώρα. Γιατί στην περίπτωση αυτή ενδεχομένω να μην μας ε, έκανε κατασκοπία η Facebook, να υπήρχε κάτι παρόμοιο. Μία ερώτηση προς τον κύριο Χάρτμαν, ο οποίος μίλησε για τον εθελούσιο χαρακτήρα που είναι επιβλαβής, γιατί ο εθελούσιος χαρακτήρας της των ε, παροχών ενδεχομένω να μην οδηγεί στο να υπάρχει το ε, ανάλογο προσωπικό για να απαντάει τα ερωτήματα αυτά. Ερωτώ λοιπόν, αν ε, ζητούμε τέτοια τεκμήρια θα πρέπει να προσλάβουν πιο πολύ προσωπικό υπάροχοι. Ποιος θα το πληρώσει, το κράτος, οι ο καταναλωτή, ποιο είναι υπεύθυνο στη χρηματοδότηση αυτών των επιπροσθέτων μέτρων. Και τον κύριο Σνάιντινγκ, να του κάνω μια ερώτηση ακόμα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των μέσων αυτών ε, των τεκμηρίων που ανέφερε. Θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ε, όπως προτείνει και ο κ. Χάρτμαν για τους δικαστές, οπότε να μην υπάρχει κοινοποίηση και να τα κοιτάει αυτά ένα δικαστή. Και ίσω ο τελευταίο ομιλητή, ο κ. Μίτσελ, θα μπορούσε να μα πει δύο λόγια. Το ανέφερε και ο κ. Μίλο πριν από λίγο, κατά πόσον είναι πραγματικά τόσο αδύνατον να χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας και κατά πόσον χρειαζόμαστε πιο πολλά στοιχεία παρά να εφαρμόσουμε το e-evidence για όλα τα εγκλήματα και θα ήθελα να ακολουθήσουμε την αντίστροφη σειρά από αυτή που ακούσαμε τους ομιλητές και να δώσω λοιπόν τον λόγο καταρχάς στον κύριο Μίτσολ για να τοποθετηθεί. Yes, the reason why... Ναι. Ο λόγος που αναφέρθηκα στην εντολή έρευνας και αυτό αναφέρεται και στο έγγραφο του οργανισμού μου. Αναφέρθηκε όμως και από άλλους ε, ομιλητές το θέμα αυτό. Αυτό διότι η εντολή αυτή υπάρχει ήδη, έχει δοκιμαστεί και δεν έχει κάποιες από τις δομικές ε, δυσκολίες και προβλήματα που έχει η νέα πρόταση. Αποτελεί λοιπόν μια κατάλληλη βάση επί της οποίας μπορούμε να χτίσουμε. Δεν θέλω να ασκήσω πολιτική και να πω τι ακριβώς χρειάζεται να αλλάξει. Γιατί αυτό συνδέεται και με το, στοιχείο, με το, με το θέμα του τι ακριβώς είναι τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Χρησιμοποιείται ο όρος αυτός, αλλά πολύ συχνά δεν κατανοείται σε βάθος. Εγώ ε, συμμετείχα και στη συγγραφή ενός ε, σχετικού βιβλίου, το οποίο είναι τόσο χοντρό, είναι τέτοιος μεγάλος ο τόμος αυτός. Πρέπει πάντως να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τα είδη του εγκλήματος που διερευνούμε και δεν είναι όλα κυβερνοεγκλήματα. Και ο κατάλογος της ε, Προεδρίας που εγώ χαιρετίζω περιλαμβάνει μια σειρά από σοβαρά εγκλήματα που δεν είναι όλα κυβερνοεγκλήματα. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το κείμενο της εντολής έρευνας, να δούμε ποια ακριβώς εγκλήματα διερευνούμε και σε ποια από όλα αυτά θα υπάρχουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, φαντάζομαι ότι θα είναι όλα τα ίδια εγκλημάτων και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το ισχύον κείμενο για την εντολή έρευνας σε ποιον βαθμό και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που επιδιώκεται με τη νέα πρόταση. Η απάντηση για μένα είναι ναι. Αν λοιπόν η απάντηση είναι ναι, τότε θα μπορούσε να τροποποιηθεί με τον δέοντα τρόπο αυτή η εντολή, η εντολή ερεύνης. Όμως ναι, δεν ξέρω αν όλοι οι συμμετέχοντες στη σημερινή συζήτηση θα ήταν έτοιμοι να εξετάσουν αυτήν την, ε, αυτό το ενδεχόμενο, αυτή την εναλλακτική. Μου φαίνεται ότι σε μια κοινωνία που βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου θα πρέπει πάντοτε κανείς να αναζητά την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση και τη χρήση υπαρχόντων συστημάτων. Γι' αυτό η CCBE θεωρεί ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να χρειαστεί ε, αυτή η εντολή διατήρησης στοιχείων. Γιατί πράγματι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα να εξαφανιστούν προτού οι διοκτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα έστω και με επιταχυμένη διαδικασία να τα ανακτήσουν. Γι' αυτό με αυτήν την εντολή, με τη διατήρηση, κανείς δεν βλάπτεται. Αν πράγματι υπάρχει ανάγκη, σε μεταγενέστερο, σε δεύτερο στάδιο, διαπιστωθεί ότι πρέπει να ερευνηθούν και αυτά τα δεδομένα. Αλλά το θέμα της εντολής υποβολής στοιχείων, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι προβληματικά. Οπότε μπορούμε, κατά τη γνώμη μας, να διατηρήσουμε ενδεχομένως ε, κάπως τροποποιημένη την εντολή διατήρησης στοιχείων και να αναθεωρήσουμε επίσης την εντολή έρευνη ώστε να ανταποκρίνεται στι ε, σημερινέ ανάγκε των διοκτικών αρχών. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε ε, χάσει ένα μισάωρο από τον αρχικό μας χρονικό προγραμματισμό, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα. Κύριε Κέρχοφ, το... τέθηκε το ερώτημα αν τα παραδείγματα που έδωσα είναι αντιπροσωπευτικά για την κατάσταση που επικρατεί. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι πραγματικά να επαναλάβω την πρόσκλησή μου και την εννοώ, είναι ειλικρινή πρόσκληση, να έρθετε στο γραφείο μου, να δείτε τους φακέλους και τις υποθέσεις που χειριζόμαστε. Για το πώς ε, λειτουργεί η αμοιβαία δικαστική σύνδρομη, να πω τα εξής. Η πρόταση το μόνο που κάνει είναι να προβλέπει να υπάρχει ένας νόμιμος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κάθε παρόχου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε δεδομένα τα οποία ε, κατέχουν πάροχοι που έχουν την έδρα τους εκτός Ένωσης. Επί της ουσίας λοιπόν όλα τα εγκλήματα, όχι μόνο τα κυβερνοεγκλήματα, διαπράττονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Τα εγκλήματα λοιπόν που διαπράττονται στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ δύσκολο να διερευνηθούν, ιδίως στο dark web. Αν λοιπόν κάποιος ε, σχημάτισε την εντύπωση ότι τα παραδείγματα που σας παρέθεσα εδώ ήταν ε, υπερβολικά, ήταν ακραία, Ειλικρινώ το λέω, ελάτε στο γραφείο μου να δείτε την κατάσταση που επικρατεί ε, και τις υποθέσεις που χειριζόμαστε. Που χειριζόμαστε. Βεβαίως η έρευνα μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα μέσα. Το να αγνοεί όμως κανείς τη σημερινή πραγματικότητα ε, είναι σαν να ε, μην έχει επαφή με την πραγματικότητα αυτή. Γι' αυτό ελάτε και δείτε και θα πιστείτε κατά τη γνώμη μου για την αναγκαιότητα αυτών των μέτρων. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, η κυρία Ιντβελτ, μα είπε ο κύριος μόλι ότι οι ευρωβουλευτέ δεν γνωρίζουν για τι πράγμα μιλάμε. Πρόεδρος, όλοι ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ίσως ε, οι συμμετέχοντες στη σημερινή συζήτηση ε, έχουν διαφορετικέ οπτικέ. Σημαντικό λοιπόν είναι να σχηματίσει κανείς τη συνολική εικόνα και όχι μόνο την μερική εικόνα της, του δικού του τομέα, του δικού του επαγγέλματος ενδεχομένω, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξουμε σε μια πολιτικά και πρακτικά ε, ορθή λύση. Γνωρίζουμε τι κάνουμε, γνωρίζουμε ποιο είναι το θέμα της συζήτησης και ταυτόχρονα όλοι μας μπορεί να μην έχουμε ε, σαφές το τι συμβαίνει στον έναν ή στον άλλον τομέα, μπορεί να μας λείπουν κάποια στοιχεία. Ο κύριος Σνάινταχαν έχει το λόγο. Θα απαντήσω εν συντομία στα γερμανικά για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας και τις δυνατότητες επιτάχυνσης των διαδικασιών. Αυτές οι δυνατότητες επιτάχυσης υπάρχουν ήδη. Αλλά απαιτείται να ε, παρεμβαίνει σε μια υπόθεση ή να χειρίζεται μια υπόθεση ένας εξειδικευμένος δικαστής που να γνωρίζει ε, τις ε, λεπτομέρειες. Αυτό βεβαίως θα, απο, θα απαιτούσε ανάλογα μέτρα από τα κράτη-μέλη, αλλά θα ήταν εφικτά. Αυτά που δεν μπορεί να καλύψει η εντολή έρευνας είναι η υποχρέωση οι πάροχοι υπηρεσιών από τρίτες χώρες να ε, ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Ένωση. Ούτε μπορεί η εντολή έρευνας να εξασφαλίσει την παροχή, την χορήγηση των δεδομένων στις διοκτικές αρχές, όπου και αν αυτά τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα. Θα μπορούσαμε βεβαίως να συζητήσουμε για μια επιταχυμένη ε, ευρωπαϊκή εντολή ε, έρευνας, αλλά θα πρέπει αυτή να ε, εξασφαλίζει το άμεσο πάγωμα των δεδομένων και τη δυνατότητά τους αυτά να υποβάλλονται σε δεύτερο στάδιο. Το άρθρο 4 παράγραφος 5 της πρότασης αναφέρει ότι αν ο πάροχος ε, θεωρεί ότι αδίκως έχει λάβει μια συγκεκριμένη εντολή, μπορεί να προσφύγει στις ε, δικαστικές αρχές της χώρας στην οποία είναι εγκατιστημένος, κάτι που μπορεί να ε, εμποδίσει σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον την υποβολή των στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Χάρτμαν. Ευχαριστώ λόγω της επαγγελματική μου εμπειρίας που κινείται στον χώρο του κυβερνητικού εγκλήματος, σας μίλησα για αυτό το θέμα, για αυτή τη διάσταση. Ξέρω όμως ότι είναι απαραίτητη η παροχή δυνατότητας 24 ώρες επαγρύπνησης από τις πλευράς των ε, διοικητικών ερχών. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις μονάδες καταπολέμησης του κυβερνού εγκλήματος, αφορά μια σειρά από ε, δικαστικές ε, μονάδες. Μπορώ, μπορεί λοιπόν να σας μιλώ εγώ από τη δική μου σκοπιά, από το δικό μου οπτικό πεδίο αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι μιλώ εκ μέρους πολλών μονάδων τμήματων των διοκτικών και δικαστικών αρχών. Σε πολλούς τομείς πλέον στη σημερινή εποχή χρειάζεται κανείς να έχει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτό αφορά δικαστικές και αστυνομικές αρχές ώστε ταχύτατα να μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις σε εξαιρετικά περίπλοκα θέματα. Στόχος μας λοιπόν είναι να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των αναγκαιοτήτων αυτών και της διαφύλαξης και της προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών. Προσπαθούμε λοιπόν τις ε, τεχνικές και επιχειρησιακές μας ανάγκες να τις συμβιβάσουμε, αν θέλετε, με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό εξασφαλίζει και αυτή η 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας μας που εξασφαλίζει την ε, σε κάθε χρόνο και στιγμή διαθεσιμότητα κάποιου δικαστικού λειτουργού προκειμένου να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε ε, παρατηρήσει βεβαίως ότι αυτή η εξειδίκευση στο δικαστικό σώμα προχωρά. Υπάρχει ε, στη Γερμανία ε, μάλιστα και εξειδικευμένο δικαστήριο κυβερνού εγκλήματος με εξειδικευμένους δικαστές οι οποίοι μπορούν να αποφαίνονται με τεκμηριωμένο τρόπο. Είπατε για, για αυτές τις ε, αντικατοπτρικές διαδικασίες. Έχουν δύο ε, διαστάσεις αυτές οι διαδικασίες. Αφενός, τα, κυβερνό, το κυβερνοεγκλήματα ε, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα τις περισσότερες φορές. Όταν λοιπόν έχω τη δυνατότητα να ζητήσω πληροφορίες και από πάροχο που έχει την έδρα του στο εξωτερικό, μου δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα να έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους μου από την ίδια χώρα ή από την άλλη χώρα, ώστε να προλάβουμε τη διάπραξη νέων εγκλημάτων. Από αυτή την άποψη είναι ένα σημαντικό ενημερωτικό εργαλείο η συγκεκριμένη έντολη. Επίσης, αποτελεί ένα εργαλείο για την απόκτηση στοιχείων σχετικά με τη διάπραξη εγκλήματος ή αξιόπινης πράξης εντός της ε, δικαιοδοσίας της χώρας, χωρίς να χρειάζεται καν δικαστική συνδρομή. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα του Τη διαδικασία έρευνας. Νομίζω ότι και τα, τα παραδείγματα που σας έδωσα εγώ και τα παραδείγματα του συναδέλφου από το Βέλγιο είναι πολύ αντιπροσωπευτικά. Και είναι αντιπροσωπευτικά για την αρμοδιότητά μου, για, την... για το κυβέρνο έγκλημα, διότι η κεντρική ε, υπηρεσία χρειάζεται να έχει εξειδίκευση, γνώσεις για την επίθεση μέσω διαδικτύου σε κρίσιμες υποδομές και τα λοιπά. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικά τα ε, δεδομένα. Για τις υποθέσεις ε, και τις απόψεις που εκφράζονται από ομοσπονδίες νομικών, δικηγόρων και δικαστών, πρέπει να σας πω ότι εγώ διαπιστώνω ότι το θέμα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων αποσχολεί πλέον ε, όλους τους κλάδους και όλες τις φάσεις της ε, δίωξης μιας αξιόπινης πράξης. Τέλος. Φυσικά, οι εμπορικές εταιρείες, χωρίς να έχω και ε, σαφή εικόνα για τις διαδικασίες της εσωτερικής αυτών των εταιρών, θα εκλάβουν αυτές τις νέες υποχρεώσεις τους ως κόστος. Είναι λογικό αυτό. Είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα στο παρελθόν ε, για το πώς ε, χειρίστηκαν οι εταιρείες αυτές τις ε, οδηγίες και τις κατευθυντήρες γραμμές που τους δώσαμε ε, για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Έγιναν επενδύσεις. Το πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθούν βεβαίως αυτές οι διαδικασίες και αυτές οι υποχρεώσεις, ε, αυτό το αφήνω στη φαντασία σας, έχω και εγώ φαντασία και μπορώ να φανταστώ κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσελ θέλει να δώσει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν. Επίσης ακούστηκε η πρόταση να αναθεωρηθεί ή να ε, ενισχυθούν μοντέλα όπως η Ευρωπαϊκή Έντολη ε, Έρευνας ε, να περιοριστεί ο ορισμός των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Όχι, με συγχωρείτε, δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Ε, γιατί έχουμε καθυστερήσει 45 λεπτά. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας. Κύριε Σνάινταχαν, εσείς έχετε πρόβλημα στη χώρα σας γιατί ζητάτε περισσότερους δικαστές. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μια, ε, ένα αίτημα δίκαιο κατά τη γνώμη μου, διότι χρειάζεται πραγματικά, πιστεύω, να επενδυθούν και να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για να βελτιωθεί η λειτουργία της δικαστικής εξουσίας. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Και προχωράμε στο επόμενο πάνελ. Μιλάμε και πάλι για τις ε, αποδείξεις σε σχέση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την αναλογικότητα και επικουρικότητα. Έχουμε λοιπόν κάποιους ακόμη προσκεκλημένους ομιλητές. Σας καλώ εδώ στο Προεδρείο. Έχουμε τον καθηγητή Μάρκο Μπόσνιακ από μέσω τηλεδιάσκεψης. Συγγνώμη που αργήσαμε τόσο πολύ και θεωρητικώς έχουμε 10 λεπτά για κάθε ομιλητή. Αν είναι δυνατόν να το μειώσετε λίγο, θα το εκτιμούσαμε όλος ιδιαίτερος. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, δεδομένου ότι περίμενε ήδη εδώ και αρκετή ώρα, σε αυτή την ε, όχι και πολύ όμορφη αίθουσα στο Στρασβούργο, θα αρχίσω δίνοντας το λόγο στον καθηγητή Μποσνιάκ. από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να μας δώσει τις απόψεις του για τις ηλεκτρονικές μαρτυρίες και ελπίζω πως θα μπορέσει να, μπορέσει να ακολουθεί την συζήτησή μας και να μας ακούει. Αν όντω ε, έτσι σημαίνει κύριε Μπόντζεκ, μπορείτε να αρχίσετε την εισήγησή σας. Ευχαριστώ και ελπίζω να με ακούτε στις Βρυξέλλες with my presentation, I was asked to do an overview of the ε, Θα σας ε, δώσω ποια είναι η άποψή μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκό Ένταλμα Υποβολή Στοιχείων ή διατήρηση στοιχείων. Είμαι δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ όμως θα σας μιλήσω ε, προσωπικά. τα πιθανές αποφάσεις ή ε, αντικατοπτρίζουν την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δει κανεί λοιπόν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παρατηρεί πως υπάρχει έλα άρθρο 8, άρθρο 13, άρθρο 6 θα εστιάσω στην παρουσίασή μου στις διατάξεις του άρθρου 8 της σύμβασης που προστατεύει τέσσερα ξεχωριστά ε, στοιχεία, δηλαδή ιδιωτική ζωή, οικογενειακή ζωή, ε, σπίτι και αλληλογραφία. Από αυτά τα τέσσερα είναι η πεποίθησή μου ότι η ιδιωτική ζωή και η αλληλογραφία είναι πρίμα φέσιε αυτά που επηρεάζονται ε, από τα προτινόμενα μέσα. Τώρα, οποιαδήποτε παρέμβαση στα δικαιώματα της σύμβασης δεν σημαίνει απαραίτητο παραβίαση των ε, λόγων δικαιωμάτων. Η αρχή του άρθρου 8 της παρέμβασης, ε, εάν γίνεται σύμφωνα με τον νόμο, εάν επιδιώκει θεμητή το στόχο και αν είναι ε, απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία μπορεί αυτά να ε, ε, εξεταστούν. Θεμητός στόχος λοιπόν, καταρχάς είναι η θέση μου ότι αυτό το κριτήριο, το κριτήριο φαίνεται να αντιστοιχεί στο προτινόμενο μέσο, δηλαδή πλήρης κατάλογος τέτοιων στόχων στη δεύτερη παράγραφο του, του άρθρου 8 της Σύμβασης περιλαμβάνει την πρόληψη του εγκλήματος στην εθνική ασφάλεια και προστασία άλλων από τα εγκλήματα αυτά. Το πρώτο κριτήριο είναι κάπως πιο επίμαχο υπό το φως των προτινόμενων μέτρων. Ε, θα... Πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει να ισχύσει αυτή η προϋπόθεση, η λόγω νομοθεσία θα πρέπει να είναι προσιτή, προβλέψιμη και να προβλέπει την προστασία ενάντια σε αυθαίρετη παρέμβαση. Στο πλαίσιο των προτινόμενων μέτρων, η σχετική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή όρια σε σχέση με την φύση του πεδίου εφαρμογή και τη διάρκεια των μέτρων αυτών, περαιτέρω τη βάση για τον, την έκδοση της ετολής, την δυνατότητα εποπτείας των μέτρων και έπειτα να οριστεί το είδος κάλυψης που προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία. Όταν μιλάμε για την απέτηση νομιμότητας, ίσως βεβαίως να υπάρξει το θέμα ε, Και έχουμε από τη μια πλευρά την προτινόμενη νομοθεσία που βεβαίως αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά υπάρχει και το θέμα του νόμου του κράτους έκδοσης και του κατά πόσο η νομοθεσία της κράτους επιβολής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όσον αφορά το νόμο του χώρας έκδοσης είναι σαφές ότι η προτινόμενη πράξη το αναφέρει σε διάφορα σημεία όπως ε, ορισμένα θέματα δεν ρυθμίζονται στην προτινόμενη πράξη όταν αναμένεται πως η αρχή έκδοσης θα εφαρμόσει διατάξεις της εγχώριας νομοθεσία. Ίσως μετά να έχουμε κάποια προβλήματα σε σχέση με αυτό, σε σχέση με την ε, το κατά πόσο είναι προσιτός και προσβάσιμος προσβάσιμη νομοθεσία της χώρας έκδοσης θα είναι σε άλλη γλώσσα μάλλον και θα αναφέρεται σε ένα αλλοδαπό νομικό σύστημα σε σχέση με την ε, προσπελασιμότητα και την προβλεψιμότητα. Αυτά όλα επιτείνονται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει απέτηση διπλής νομιμότητας στον προτινόμενο κανονισμό, ούτε υπάρχει ένας κανόνας, κατάλογο συγγνώμη, ε, αδικημάτων, πράγμα που σημαίνει μεγάλη διαφορά από άλλα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, για παράδειγμα. Επιπλέον δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την ύπαρξη ή παρόμοιων μέτρων στο σύστημα του κράτους επιβολής. Δηλαδή ένα μέτρο μπορεί να ε, πρέπει να ληφθεί, ενώ δεν υπάρχει στο νομικό οπλοστάσιο του κράτους επιβολής. Βέβαια, όλοι αναμένεται να γνωρίζουν το χώριο δίκαιο της λόγω χώρας και το ευρωκοινοτικό δίκαιο, αλλά δεν με αν κανείς μπορεί να είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει την ε, ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους μέλους της Ένωσης. Όσον αφορά το κράτος επιβολής, φαίνεται να μην έχει σχέση με, για την ε, εν λόγω πρόταση. Τώρα, για ένα κομμάτι της σύμβασης αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα γιατί Έχουμε 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπογράφουν την ε, σύμβαση και τα οποία είναι υπεύθυνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δική τους επικρότεια και δικαιοδοσία. Θα πρέπει να θεσπίσουν νομικό πλαίσιο και να εγγυηθούν νομική και δικαστική προστασία ακόμα σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει στο παρελθόν ασχοληθεί με υποθέσει αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή έχει δεχτεί την, το τεκμήριο της ίσης προστασίας, όμως εάν οι αρχές της χώρας επιβολής αντιμετωπίσουν καταγγελία ότι η προστασία των συμβατικών δικαιωμάτων είναι ελλειπής και ότι αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, θα πρέπει να εξετάσουν την καταγγελία επί τη βάση του ότι απλώς εφαρμόζουν την ε, κοινωτική νομοθεσία και αυτό έχει σαφώς δηλωθεί στην απόφασή μας ΑΟΚΙΝΣ εναντί Λετωνίας και έχει επικυρωθεί επανελειμμένα. Η πρόταση είναι αρκετά μοναδική όσον αφορά την ομολογία ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή η η, παρέμβαση του άρθρου 8 δεν μπορεί να επιβληθεί. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί μπορεί να υπάρχει μια θεμητή προσδοκία ότι το, το οικείο δίκαιο θα εφαρμοστεί κάθε φορά. Simply Add the proposed and Τώρα, αν έχουμε μια κατάσταση στην οποία θέλουμε να αξιολογήσουμε από την άποψη της απέτηση του δικαίου του ίδιου και να δούμε κατά πόσο οι διατάξεις του παρέχουν αποτελεσματικές εγγύησεις κατά κατάχρησης υπό, υπό το φως της ε, νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Το πρώτο ζήτημα είναι κατά πόσο το περιεχόμενο των προβλεπόμενων μέτρων είναι επαρκώς ορισμένο. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν είμαι ειδικός για κάποια θέματα τεχνολογίας, ωστόσο φαίνεται πως κάποιες φορές είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κατά πόσο ένα συγκεκριμένο μέτρο ή ένα συγκεκριμένο βήμα η εντολή για την υποβολή στοιχείων πρόσβασης, στοιχείων συνδρομητή ή στοιχείων συναλλαγών ή οτιδήποτε παρόμοιο. Ας πούμε, Εάν δούμε την υπόθεση Μπενέντικ έναντι Σλοβενίας που αναφέρθηκε από κάποιον από τους προηγούμενους ομολητές, μπορεί όντως εκεί να μην ήταν ξεκάθαρη η υπόθεση. Επιπλέον δεν γίνεται αναφορά στην πρόταση για το περίοδο και τη διάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων, τη διαδικασία κύρωσης, η οποία δεν περιγράφεται πολύ σαφώς, δεν υπάρχουν διατάξεις για την εποπτεία της διαδικασίας και την εφαρμογή των μέτρων και υπάρχουν περιορισμένες διατάξεις για τις διαθέσιμες νομικές καλύψεις. εφόσον ε, δεν θα υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένες διατάξεις για τα κριτήρια, όταν κανείς εξετάζει αυτή την πρόταση, να πω συνολικά και σύντομα θα σταθώ στο θέμα της σοβαρότητας του αδικήματος, όπου η, εντολή, η ευρωπαϊκή εντολή υποβολής δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει για όλες τις, ε, ταπεινικά δικήματα ε, για τουλάχιστον τρία χρόνια. Για, σύμφωνα με ορισμένα νομικά συστήματα, πολλά δικήματα εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Διαταγή ένταλμα μάλλον διατήρηση αφορά όλα τα δικήματα και δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά την απόδειξη και δεν υπάρχουν όρια για τη διάρκεια του μέτρου και την μετέπειτα χρήση των ε, δεδομένων που έχουν αποκτηθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω αυτή η ε, πρόταση ε, και φυσικά ευχαρίστως να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να σου το λόγο παρά αυτά στον επόμενο μαγητή, ο οποίος είναι ο κύριος Τιρίνγκ. Ο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε τη λόγο. Έχουμε πολλά ακούσει ήδη από τους εμπειρογνώμονες και δεν χρειάζεται να επαναλάβω πολλά εξ αυτών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους συμμετέχοντε ότι στην αρχή ο κύριος Μπέος κατέστησε σαφέ ότι υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά στην Ομίγυρη για το θέμα της ε, επικυριαρχίας, της ε, δικαστικής προστασίας. Αυτό καθίσταται όλο και πιο σαφέ, σαφές από αυτά που είπε και ο κ. Μπόσνεκ. Η επικυριαρχία σημαίνει ότι όλες οι χώρες που έχουν προσυπογράψει την ε, χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα δεσμεύονται να εξασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα στην επικρατεία τους. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η πρόταση αυτή τηρεί την αρχή αυτή επιτρέποντας τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο εποπτείας. Το άλλο θέμα είναι η δικαστική αναθεώρηση, ο δυστικός έλεγχος. Εδώ υπάρχουν κάποια κενά τα οποία μπορούν να πληρωθούν. Θα αναφέρω κάποια εξ αυτών. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπαν οι προλαλήσαντες και κυρίως ο κύριος Μπέος, ο κύριος Νέντραχαν και ο κύριος ε, Βασίκα. Υπάρχει ο, ο σε μια τέτοια κατάσταση να παραβλέψουμε άλλου κίνδυνου, άλλα προβλήματα και θα ήθελα να θέσω και κάποια ίσονο σημασία σε προβλήματα τα οποία παρόλα αυτά έχουν να κάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο άρθρο 2 υπαριθμό 15 εδώ ορίζονται οι περιπτώσεις κατεπίγουσας ανάγκης. Το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να περιορίσουμε αυτές τις περιπτώσεις σε απειλές για τη ζωή. Για παράδειγμα, οι προσβολές στην αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου δεν, καλύπτουν, δεν καλύπτονται από απειλές στη ζωή τους, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ή, για παράδειγμα, αν προγραμματίζεται απαγωγή ενός ατόμου, αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα ε, απειλή στην σωματική ακαιρεότητα ενός ατόμου, ένα παιδί για παράδειγμα, πρέπει να, να προστατεύεται από τη σεξουαλική πορνογραφία. Άρα ο ορισμός για το τι αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη στο 2015 είναι πολύ περιορισμός. Θα πρέπει να παρέχεται προστασία σε οποιαδήποτε πράξη που απειλεί άμεσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια βάσει του άρθρου 1 της χάρτας και ο 2 έως 7 άρθρα του χάρ, της χάρτας. Μία ερώτηση για το άρθρο 5. Σε ό,τι αφορά την σειρά παραγωγή, στο άρθρο 5, παραγραφός 4, ορίζονται τα δικήματα για τα οποία μία εντολή μπορεί να εκδοθεί σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα ιδεχθείς, ε, ιδιαίτερα μεγάλα δικαιώματα. Βασιζόμαστε στη μέγιστη ποινή. Ωστόσο, η ακρίβεια του μέτρου αυτού είναι αμφισβητήσιμη. Ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 9, 25 κράτη-μέλη υποχρεούνται να ποινικοποιήσουν ε, την ε, κατάχρηση εργαζομένων από τρίτες χώρες σε ακραίες συνθήκες εργασίας. Και αυτό συνεπάγεται κάθε 6-5 ετών. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η ποινή είναι 2-5 χρόνια. Για το Λουξεμβούργο όμως αυτό συνοδεύεται με φυλάκιση 8 ε, μήνες, 8 μέρες έως ένα μήνα. Στην Τσεχική Δημοκρατία αυτό ανέρχεται στους 8 μήνες, η φυλάκιση ανέρχεται στους 8 μήνες. Άρα αυτό που αποτελεί σοβαρό αδίκημα σε μια χώρα είναι πιο ίσονος ε, σημασία ε, σε άλλη χώρα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν και σοβαρά εγκλήματα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην κατηγορία σοβαρών εγκλημάτων, όπως ορίζεται στον κανονισμό της Europol. Και συμπεριλαμβάνονται μια μεγάλος κατάλογος ε, αδικημάτων. Επίσης, 5-4β. Στο άρθρο 5-4β αναφέρονται διάφορα αδικήματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται γιατί ε, διαπράττονται μέσω συστήματος επικοινωνίας, για παράδειγμα ε, παραχάραξη online πληρωμών, πατική πορνογραφία και ούτω καθεξής. Αυτό που θα πρέπει να προσταθεί είναι τα εγκλήματα ε, μίσου online σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση ρατσισμού, ξενοφοβίας. Τα κράτη-μέλη άλλωστε υποχρεούνται να ποινικοποιούν τέτοιε μορφές βίας. Στο Αθενέ, παράγραφος 2, του πλαισίου απόφαση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία περιλαμβάνει υποθέσει όπου η συμπεριφορά γίνεται μέσω συστημάτων online. Το θέμα των, της παρότρινσης εμίσους αποτελεί ένα άλλο και ε, αυξανόμενο φαινόμενο. Και αυτό οδηγεί σε ξενοφοβικές ε, τάσεις. Είναι πολύ σοβαρό και να στραφώ στο άρθρο 14. Μια γενική παρατηρήση καταρχά. Όποτε η πρόταση αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα, φαίνεται λε και περιορίζουν την δράση των αρχών. Είναι το κράτος ενάντια του κατηγορούμενου, του αναγόμενου. τα δικαιώματα του πολίτη και του κατηγορούμενου επηρεάζονται από τα συστήματα. Αυτός που δεν εμφανίζεται στο μοντέλο αυτό όμως είναι το θύμα. Και αυτό το σύστημα δικαστικής αγωγής ε, έχει σιγά σιγά παροχηθεί και αναδείται ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο μηχανισμό ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, ατόμων, των θυμάτων. Αναγνωρίζεται ότι τα σοβαρά εγκλήματα αποτελούν σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άρα τα θύματα τέτοιων παραβιάσεων έχουν δικαίωμα να κάνουν αγωγή, ποινική αγωγή, ως η μοναδική αρμόζουσα ένομη λύση σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων του εκάστοτε θύματος. Τα θύματα λοιπόν τέτοιων εγκλημάτων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποτελεσματική έρευνα για την εντοπισμό και την τιμωρήση των ε, υπετίων και Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι μια υπόθεση της Φιλανδίας από το δικαστήριο στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι αρχές έχουν όλα τα εργαλεία για να εντοπίζουν και να καταδικάζουν τους υπετίους. Ε, και ό,τι προκύπτει από τον κανονισμό ως υποχρέωση θα πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, θεμάτων Και αυτό με φέρνει στο άρθρο 14 της πρότασης. Ένα βασικό στοιχείο της έκθεσης είναι η αναγνώριση της ε, εντολής. Ωστόσο, στο θέμα αυτό, εδώ η πρόταση μας δίνει αντικρουόμενα μηνύματα. Ένα σημείο αναφέρεται στην παραγραφό 2 ότι οι αρχές αναγνωρίζουν μια εντολή χωρίς περαιτέρω τυπικές διαδικασίες. Από την άλλη, στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι οι αρχές επιβολής θα πάρουν την απόφαση να αναγνωρίσουν την ε, εντολή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της ε, εντολής. Άρα, ποιος είναι τελικά αυτός τον οποίο απευθύνεται ο καθού της ε, εντολής. Η μοναδική λογική απάντηση είναι ότι η απόφαση αυτή απευθύνεται στον εκάστοτε πάροχο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, στο 14.2, και το 14.3 ζητούν να συνάδει ο πάροχος με τις σχετικές υποχρέωσεις. Αυτό που φαίνεται σαν δύο βήματα της ίδιας διαδικασίας, αναγνώριση της ε, εντολής και απόφαση να συμμορφωθούν ε, τελικά με τις ε, διατάξεις. Αυτό είναι ουσιαστικά μία απόφαση και αν είναι η απόφαση αυτή δεσμευτική και επηρεάζει λοιπόν την ε, ελευθερία διεξαγωγής συναλλαγών υπό το άρθρο 6 του χάρτη και του και έτσι θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 47 του χάρτη του μελετών δικαιωμάτων, υπάρχει δυνατότητα αγωγή έναντι τη απόφαση αυτή από πλευρά του κατηγορούμενου. Και φαίνεται ότι πάλι η αρχή εφαρμογή είναι αυτή που πρέπει να έρθει σε επαφή με τον πάροχο. Αυτό όμω δεν αποτελεί πραγματικά νόμο μέσω βάση τη άρθρου 47. Να θυμόμαστε ότι οι αρχέ του κράτου μέλου θα δρεύουν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου και έτσι ισχύει ο χάρτης των δικαιωμάτων. Θα έχουν δηλαδή τέτοια ζητήματα Θα πρέπει να υπάρχει ενδικό μέσο υπό την έννοια του άρθρου 47 του χάρτη, ένα ανεξάρτητο δικαστήριο δικαιώματα για δίκαια δίκη και την ε, διαθεσιμότητα νομικών πράξεων. Η πρόταση λοιπόν δημιουργεί μια διτότητα με ένα παράλληλο χαρακτήρα μεταξύ των εντολών που εκδίδονται από την αρχή έκδοση και αποφάσει που λαμβάνονται από την αρχή εφαρμογή για την αναγνώριση των εντολών αυτών. Θα είμαι σύντομος, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι η αναγνώριση της ε, απόφασης θα πρέπει να γίνει βάσει των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και 5 στο άρθρο 14, παράγραφος 4 και 5. Ένας ε, μακρύς κατάλογος ότι έχει εκδοθεί, έχει επαληθευτεί η εντολή. Στο άρθρο 5 θα θυμάστε ότι τα κριτήρια είναι αρκετά ακριβή. Αν η αρχή εφαρμογή χρειάζεται να ερευνήσει όλες αυτές τις ε, προαπαιτήσεις πρωτού αναγνωρίσει την εντολή, εδώ βασιζόμαστε στις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης. Είναι βασικά στοιχεία αυτά όμως για την αποτελεσματικότητα της έρευνας σε διασυνοριακές καταστάσεις. Η δικαιολόγηση της πρότασης έχει να κάνει με την ναι, σα, ε, σημαντικό κέρδο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα. Αλλά όσο αφήνουμε έξω τις αρμοδιότητες του κράτους έκδοση, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουμε σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα. Και αυτό σημαίνει ότι χάνουμε ό,τι κερδίζουμε σε αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο απευθείας στον επόμενο προσκεκλημένο ομιλητή, τον κύριο Μακναμή από την Έντρη. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Σε αυτήν την εξαιρετική ε, συζήτηση με τους εξαιρετικούς συμμετέχοντες που έχουν αναφερθεί σε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς την ε, Επιτροπή σας για τα ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος ε, δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που έχουν ανακύψει σε μια σειρά από κράτη-μέλη. Χθες το Ευρωβαρόμετρο ε, αποκάλυψε, διαπίστωσε ότι ε, σε 9 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση της δικαιοσύνης και της δικαστικής εξουσίας σε γέννη. Αυτό ε, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη σε μια περίοδο που είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Θέλω να επικεντρωθώ, να επικεντρωθώ στο ποιο είναι το νόημα της πρότασης. Αν είναι η λιγότερο περιοριστική εναλλακτική, αν ε, σέβεται τις νομικές διαδικασίες, ε, αν εξασφαλίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μιλών για ισορροπία και ποια είναι η απάντηση που μπορεί να δοθεί στους, ε, στις νομικές αμφιβολίες που εξέφρασε και ο δικαστής Μπόσνακ πριν από λίγο. Ο δικαστής λοιπόν έθεσε το ζήτημα της νομικής προβλεψιμότητας. Ακόμη και αν όλα τα άλλα μείνουν ίδια, στις πλέον ε, σημαντικές προτάσεις αν η ε, κατάσταση αλλάξει σε μία από τις ε, νομοθεσίες τότε τα πράγματα γίνονται προβληματικά. Είναι η λιγότερο παρεμβατική εναλλακτική. Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η, απόδοση, η απονομή δικαιοσύνη είναι αργή. Όμως είναι λογικό σφάλμα και άλμα να πούμε ότι επειδή κάτι δεν έχει λειτουργήσει, δεν μπορεί και να λειτουργήσει στο μέλλον. Η Κομισιόν έκανε πολύ καλή δουλειά στην έκθεση προόδου και ε, προσδιορίσε τις ε, όριμες δυνατότητες που υπάρχουν για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας. Βεβαίω, αν χρησιμοποιούμε αυτό τον σύντομο δρόμο, ποιο θα κάτσει να κάνει τον μεγάλο δρόμο. Παρομοίω, η ΕΠΑ ε, εισήγαγαν μια μεταρρύθμιση του ΕΜΛΑΤ που μείωσαν τη συσσόρευση ε, δικαστικών υποθέσεων κατά το 1 τρίτο αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι το γεγονός ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου χρονικού δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και στο μέλλον. Ε, η, Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε ε, στο παρελθόν την Ευρωπαϊκή Έντολη Έρευνας χωρίς να έχει ακόμη κατά νου τα, τα ψηφιακά δεδομένα. Τώρα ξαφνικά ε, φαίνεται να επανέρχεται με μεγαλύτερη επιτακτικότητα αυτή η διάσταση των ψηφιακών δεδομένων. Επίσης, το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών. Το κράτος έκδοσης πρέπει να σέβεται τις ε, νομικές ε, υποχρεώσεις και εγγυήσεις που υπάρχουν στη χώρα ε, παραλαβής της εντολής. Αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει ε, η δικαστική, εξουσία, η δικαστική αρχή της χώρας έκδοσης να σέβεται την ένωμη τάξη μιας άλλης χώρας προσπαθώντας να μην την παραβιάσει. Ε, εκφράζω την αμφιβολία μου για το αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Οι δικαστικές δε αρχές του κράτους παραλαβής ε, της εντολής θα ενημερώνονται μόνο σε περίπτωση καταγγελίας του παρόχου. και εκείνο θα πρέπει να επικαλείται σοβαρή και εμφανής παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όχι μόνο δηλαδή να είναι σοβαρή, να είναι και εμφανής και να εκδηλώνεται με αυτό τρόπο. Άρα ο ε, δικηγόρος της εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και στοιχεία ε, του μη εταιρικού δικαίου για να μπορέσει να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη γνώμη για να προβεί στην, στο παράπονο, στην καταγγελία. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα τεκμηριώσει ο πάροχος στις τέσσερις σελίδες στις οποίες έχει στη διάθεσή του για να ε, υποβάλει την ένστασή του. και ταυτόχρονα, αν εκτελέσουν την εντολή, τότε δεν διατρέχουν κίνδυνο. Αν όμως υποβάλουν ε, καταγγελία, αν υποβάλουν ένσταση, τότε ε, είναι αντιμέτωποι με ε, πρόστιμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ανισο, ανισορροπίας των κινήτρων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε αποφανθεί σε άλλη υπόθεση ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ε, εξασφαλίζουν τη ισορροπία του ενωσιακού δικαίου, της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου με, το, με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, πολιτών τους. Είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν ε, εξαίρεση για τους ε, παρόχους που λειτουργούν καλή την πίστη, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των πελατών τους. Άρα, αν κάποιος πάροχος λάβει μια τέτοια εντολή, μπορεί πάντοτε να ισχυριστεί ότι ε, ενεργούσε καλή την πίστη. Δεν ενημερώνεται λοιπόν ο ενδιαφερόμενος, δεν, ενδιαφερόν, δεν ενημερώνεται το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το κράτος μέλος υποδοχής αυτής της εντολής και, δεν, και ταυτόχρονα μπορούν και να επιβληθούν πρόστιμα σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί κανείς. Αυτό δεν ε, θα το χαρακτήριζα ισορροπημένη πρόταση. Η συλλογή μεταδεδομένων ε, μπορεί να είναι εξίσου παρεμβατική με τη συλλογή δεδομένων περιεχομένων. Έχουμε λοιπόν αμφιβολία όσον αφορά την ε, συμμόρφωση αυτής της πρότασης με την ομολογία του δικαστηρίου σε διάφορες υποθέσεις που αναφέρθηκαν. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο ε, χτίζονται πολιτικοί συμβιβασμοί γύρω από αμφιλεγόμενους ορισμούς που αφορούν κυρίως τα μεταδεδομένα. Μπορεί να βασίζονται σε κάποιες πολιτικές αρχές, οι οποίες όμως δεν μπορεί να αναιρέσουν βασικές νομικές αρχές. Και μετά ε, μιλάμε για την επιλογή του, της νομικής πράξης. Επελέγει ο κανονισμός. Ενδιαφέρον αυτό, διότι Τέθηκε και το ερώτημα αν πρακτικά είναι κάτι τέτοιο εφαρμόσιμο. Τι σημαίνει όμως, γνωρίζουμε από το ιστορικό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, απέρριψε το, την πρόταση περί ασφαλούς λιμένα παρά την νομική ανάλυση στην οποία έχει προβεί η Κομισιόν, όπως επίσης απέρριψε και το PNR Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, παρά την αντίθετη ε, νομική ανάλυση της Κομισιόν. Δεν αποκλείεται να συμβεί το ίδιο και, και με αυτές τις προτάσεις που υπέβαλε τώρα η Κομισιόν. Τι θα γίνει λοιπόν αν επαναληφθεί η ιστορία. Αν εγκριθεί αυτός ο κανονισμός και τεθεί σε εφαρμογή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάνει ακριβώς αυτό που είχε κάνει και με την ε, οδηγία για την διατήρηση των δεδομένων. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Το να, εγκρι... το να εγκριθεί δηλαδή μια νομική πράξη η οποία δεν θα ευσταθεί και θα καταρριφθεί με την πρώτη ευκαιρία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομίζω ότι πλήττει σοβαρά το κύρος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Εμείς υποστηρίζουμε τα θεμέλια της δημοκρατικής μας κοινωνίας όπως αυτά καθορίζονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει η πρόταση είτε να τροποποιηθεί σημαντικά είτε να αποσυρθεί. Να προσδιοριστεί καταρχάς ε, να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να, να βελτιωθεί η εντολή έρευνας και να διευρυνθούν οι εγγυήσει και να επιλέγεται πάντοτε ο λιγότερο παρεμβατικός τρόπος, η λιγότερο παρεμβατική εναλλακτική. Επίσης, απαιτούμε να διαφάνεια όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται για το παράρτημα της σύμβασης ε, Cybercom. Εσείς ως εισηγήτρια γνωρίζετε τα θέματα αυτά, τα αυτά είστε ευαισθητοποιημένοι. Ε, το ίδιο και η στάση των 8 κρατών μελών που έχουν εκφράσει αμφιβολίες. Χαιρετίζουμε και την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και <clears throat> προσβλέπω και στην ε, συνεργασία στη συνέχεια μαζί σας. Σας ευχαριστώ και ελπίζω όλοι οι παραγοντάς στη διαδικασία αυτή να έχουν ε, ε, συμφέρει να δημιουργήσουν μια νομοθεσία η οποία θα στέκει. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την πληροφορία αυτή, για τις πληροφορίες αυτές. και τον κύριο Πόσνιακ από το δικαστήριο παρά το γεγονό ότι σημείωσε ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Θα τα λάβουμε φυσικά αυτό υπόψη. Επόμενο ε, Ομιλητή ο κύριο Βιβιερόφσκι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία Δεδομένων. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά και ευχαριστώ πάρα πολύ και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο μια και τα πιο πολλά στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί από του προηγούμενου ομιλητέ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ και συνεισηγητέ, αγαπητέρνοι προσκεκλημένοι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω καταρχά για την πρόσκλησή σα εδώ για να παρουσιάσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων που λαμβάνει μέρος και στην ε, αρχές ε, προστασίας δεδομένων στο Συμβουλίο, Συμβούλιο. και στη Σχετική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι κατανοούμε απόλυτα ότι σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος διαρκώς και συνεχώς βρίσκεται υπό μεταλλαγή από τις νέες τεχνολογίες. Με χαρά μας χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά εκ παραλλήλου θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι εγκληματικές δραστηριότητε επίσης έχουν ωφεληθεί από αυτές τις νέες οδούς δράσης και προκύπτει από τα αποδεκτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις εγκληματικές αυτές ενέργειες ότι συχνά αυτά εντοπίζονται σε επίπεδο ηλεκτρονικό. Είναι δύσκολο να φανταστούμε μια ποινική έρευνα που δεν θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά τεκμήρια. ή αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Να καταλάβουμε λοιπόν. Αυτό ήταν σαφές από την παρουσίαση του κ. Κερκόφ. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνει ότι δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε καμία αρμοδιότητα από τις αρχές και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε λέιζερ προς την κατεύθυνση αυτή. Ήθελα ωστόσο να είμαι ξεκάθαρος. Ο Ευρωπαϊκός Επόπτης για τα δεδομένα κατανοεί και υποστηρίζει το στόχο να παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία στις ε, αρχές επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Θα είναι καινούργια όμως αυτά τα εργαλεία ή είναι αυτά που χρησιμοποίησαμε το 2014 και ακόμα δεν έχουν ε, εφαρμοστεί πλήρως και δεν έχει μάλλον αναφερθεί κατά πόσον είναι αποτελεσματικά ή όχι. Επίσης, η πρόσβαση στα τεκμήρια αποτελεί μία από τις εκ των ουκάνεφε προϋποθέσεις για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς. Αυτό δεν είναι καθε αυτό αντίθετο με την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δημιουργούμε μια τέτοια αντίφαση μεταξύ της πρόσβασης ε, στα τεκμηρία αυτά και της προστασίας των δεδομένων. Δεν υπάρχει κάτι το καινούργιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης. Αυτό που είναι καινούργιο στην πρόταση είναι η διασυνοριακή διάσταση. Αυτό είναι το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές της πρώτης χώρας μπορούν να ζητήσουν πιο γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα μιας δεύτερης χώρας χωρίς να περνάνε μια μακρά διαδικασία. Και πιστεύουμε ότι είναι βασική σημασία να διευκρινιστεί στο νομικό κείμενο ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι νέοι ουσιαστικά. Επίσης, αυτή η νομοθεσία θέλει ουσιαστικά να εφαρμόσει αρχές που ήδη υφίστανται. στοιχεία που έχουν ήδη εφαρμοστεί από το Κοινοβουλίο, έχουν ήδη περάσει από το Κοινοβούλιο το 2016 και εφαρμόζονται. Ενδεχομένω να υπάρχουν αμφιβολίε για το πώ εφαρμόζονται, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία για να ελέγξει το πώς το πετυχαίνουν αυτό τα κρατη Είναι λοιπόν βασικό να διατηρηθεί αυτός ο σύνδεσμο μεταξύ της και των αρχών επιβολής του νόμου. Ωστόσο, αν η προτινόμενη νομοθεσία έχει να κάνει μόνο με τους τρόπους διατύπωσης ε, υφιστάμενων ε, αρχών, να διευκρινίσουμε ότι ακόμα και ε, αυτές έχουν ε, ενδεχομένω συνέπειε σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι ε, θεμελιώδει ελευθερίε. Και αυτό πιστεύουμε ότι ισχύει στην πρόταση αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε σύντομα σε θέση να προτείνουμε συγκεκριμένε τροπολογίε για να περιοριστεί ο παράπλευρε απόλυε, αν θέλετε, σε σχέση με την πρόταση. Και γι' αυτό χάρηκα με την παρουσίαση του καθηγητή Πόσνεκ. Και μια και η νομολογία του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί τη βάση για τις ε, αρχές επιβολής του νόμου. Αλλά και πιο σημαντικό για τις μεμονωμένες, ε, τα μεμονωμένα 11 μέσα που παρέχονται στο κάθε κατηγορούμενο. Η αρχές προστασίας των δεδομένων περιλαμβανομένου και του EDPS ε, έχουν ήδη εκδώσει την γνωμοδότησή τους για την ε, πρόταση αυτή. Η πρότασή μας θα συμπληρώσει την γνωμοδότηση αυτή. Τώρα θα ήθελα να διευρύνω το πεδίο των σχολείων μου, των παρτρήσεων μου και να κοιτάξουμε λίγο πιο πολύ την ευρύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τεκμήρια. Όπως γνωρίζετε, οι συζητήσει για το δεύτερο συμπληρωματικό πρωτόκολλο για το κύβερνο έγκλαμα είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των αρχών να συνεργάζονται άμεσα με τους παρόχους ε, των άλλων δικαιοδοσιών. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τις συζητήσεις αυτές με προσοχή και τις εξελίξεις που θα σημειωθούν και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, θέλει να αρχίσει τις συζητήσεις σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τεκμήρια με τις ΕΙΠΑ, αλλά να σας διευκρινίσω ότι αυτή η πρόταση δεν περιλαμβάνει αυτό. Ακούμε ότι μας δίνει τα εργαλεία να επιλύσουμε το θέμα της πρόσβασης ε, των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στι ΕΙΠΑ. Και αυτό δυστυχώ ε, μου υπενθυμίζει ότι ό,τι απόφαση και να λάβουμε εδώ σε αυτήν την αίθουσα, αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα και θα πρέπει να σκεφτούμε και τα επόμενα βήματα. Να σκεφτούμε λοιπόν τις προτάσεις αυτές, να έχουμε υπόψη μας και το μέλλον. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι της όλης της ιστορίας. Και εδώ κατανοούμε ότι η συζήτηση αυτή θα μας ε, απασχολήσει τα επόμενα δύο έτη. Το κλειδί για την εξασφάλιση ότι το τελικό κείμενο θα εξασφαλίζει πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και δεν θα αποκλίνει από το εφιστάμενο πλαίσιο. Θα ήθελα να αναφέρω και άλλο ένα κομμάτι νομοθεσία, άλλο ένα νομοθετική πράξη που συνδέεται με αυτά το, το θέμα. Οι αποφάσει και συστάσει του Ευρωπαϊκού Επόπτη Δεδομένων θα πάνε χέρι-χέρι με τις προτάσεις για την τρομοκρατία γιατί υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Όπως έχει σημειωθεί για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια εδώ, σε αυτό το φάκελο, δεν υπάρχει κανένα σημαντικό ζήτημα. Είναι δυνατόν να βρεθεί συμβιβασμό από αυτού. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξή. Δεδομένων των, της σημασίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά πυρνικά ζητήματα. Και ρεαλιστικά θα μας πάρει κάποια χρόνια να αναγνωρίσουμε όλα τα σημαντικά γεγονότα του κανονισμού. Παρ' όλα αυτά, η συνοχή με το εφιστάμενο πλαίσιο προστασίας δεδομένων θα πρέπει να ιδρυθεί Και οποιαδήποτε αντίληψη απόκληση από το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία στη μελλοντική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, λέει και η Πρόεδρος, για την παρουσίαση αυτή και ασφαλώς. Όλα τα πάνελ έχουν επαναλάβει κάποια πράγματα, αλλά βρίσκουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα σημεία αυτά που προέκυψαν σε όλα τα πάνελ, ότι δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες έχουν πολλά στοιχεία στις ΕΠΑ, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, όπως εγώ ερμηνεύω αυτά που είπατε, είναι μήπως θα έπρεπε πάνω απ' όλα να σκεφτούμε συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να αγκάσουμε όλους να το αντιμετωπίσουν. Τώρα προχωρούμε προς το τέλος αυτού του πάνελ και με τα χαράς ε, θα δώσω το λόγο στον ε, ομιλητή από στην ομιλήτρια από την Εθνική Επιτροπή Πληροφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Μπρουνέ, έχετε το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Πολλά από τα σημεία που ήθελα να αναφέρω αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων τον περασμένο Σεπτέμβριο υιοθέτησε και δημοσίευσε την θέση της και τις προτάσεις της για το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς να σας παρουσιάσω τις ε, σειρές παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή τη γνωμοδότηση και έπειτα τις πιο λεπτομερείς αναλύσεις και εγγυήσεις που έχουμε παρατηρήσει ή των οποίων η έλλειψη μας εντυπωσίασε μέσα στο πλαίσιο των ε, διαδικασιών έκδοσης ενταλμάτων. Προστασία δεδομένων, ε, πρώτη σειρά παρατηρήσεων ε, αφορά την νομική βάση, δεν χρειάζεται να επανέλθει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασία Δεδομένων ε, έχει εκφράσει τις ίδιες αμφιβολίες για την νομική βάση που αφορά την δικαστική εγγύηση όταν ένα από τα, από διάδικα μέρη είναι ιδιώτης. Η Επιτροπή εξέδασε την ανάγκη ύπαρξη αυτής, ε, αυτού του μέσου σε σχέση με τις συμφωνίες δικαστικής αρρωγής και ε, ε, διέβλεψε ότι υπάρχουν λίγα μέσα εκεί υπάρχει έλλειψη εναλλακτικών ε, προτάσεων για να βελτιωθούν τα ήδη υπάρχοντα μέσα, τα οποία θα μπορούσαν και να αρκέσουν. Εξετάσαμε και τις συνέπειες σε θέματα εγγύησης και προστασίας των δεδομένων ε, των ενδιαφερομένων ε, ατόμων όταν πρόκειται για την εγκατάλειψη της αρχής της διπλής απαγγελίας κατηγορίας που διαπιστώνουμε ότι σε θέματα ποινική διαδικασία προβλέπονται κάποιες εγγυήσεις και από την άποψη της προστασίας των δεδομένων δεδομένων, ορισμένε από τι εγγυήσει τη ποινική διαδικασία ακριβώ αυτό θέλουν να εγγυηθούν, την προστασία των ε, διαδίκων και η φόβη μας είναι η εγκατάλειψη αυτού του διαλόγου για αυτό το θέμα και αυτών των επιπλέον εγγύησεων. Τέλος, τελευταία σειρά παρατηρήσεων σε σχέση με την ανάγκη αυτών των νέων μέσων, ε, ε, εξετάσαμε τις συνέπειες της αντικατάστασης ενός από τους συνομιλητές στο διάλογο, που δεν είναι πια μια δικαστική αρχή, αλλά αποτελεί και μετατρέπεται σε ιδιότητα. Ε, ε, άρα λοιπόν το βάρος το οποίο θα πρέπει να φέρουν αυτές οι εταιρείε για να εγγυηθούν το σεβασμό των δικαιω... θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί ένας από τους στόχους ε, των δικαστικούς είναι να εγγυηθούμε μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων και γενικών αρχών του κράτους δικαίου που θεωρούμε πως είναι μια δυσανάλογη αποστολή για ιδιώτες φορείς που επιδιώκουν άλλους στόχους και όχι την προστασία του κοινού συμφέροντος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι αρχές της προστασίας δεδομένων. Έτσι αυτές οι αρχές μπορούν και πρέπει να επιβλέπουν την εξέλιξη και την εκτήληξη της διαδικασίας και αυτές θα έπρεπε να εγγυηθούν το γενικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. Troisième série de remarques générales que nous formulons, et c'est directement lié à ce, ce que je viens de mentionner, euh, c'est l'applicabilité des garanties. <laughs> εφαρμογή των εγγυήσεων, ή είναι οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο ποινικό τομέα και ιδιαίτερα το άρθρο 39 ε, για θέματα μεταφοράς δεδομένων και διαλόγου ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές στις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικών φορέων, εκτός της Ένωσης δηλαδή. Αυτές οι εγγυήσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν σε τέτοιου είδους περιστάσεις ε, συγκεκριμένα και θεωρήσαμε απαραίτητο ότι, ε, να θυμίσουμε ότι αυτό το άρθρο πρέπει να εφαρμόζεται και πρέπει να υπάρχει και μια τεκμηρίωση για μεταφορά των δεδομένων όταν αυτά, αυτή η μεταφορά γίνεται. Και έπειτα μετά από αμοιβαίο αίτημα, εφαρμογή του άρθρου 48 του Γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων που προβλέπει εγγυήσει όταν στοιχεία Ευρωπαίων ζητώνται από αρμόδιες αρχέ εκτό Ένωση. Και η τελευταία σειρά των γενικών παρατηρήσεων θα πρέπει να διευκρινιστεί γιατί ακριβώς αντικατοπτρίζει παρόμοιες έννοιες σε άλλα μέσα όπως είναι η έννοια του παρόχου υπηρεσιών, των ε, ε, επιχειρήσεων, ε, ομίλων επιχειρήσεων που καμιά φορά ομαδοποιούν αυτά τα θέματα της ε, προστασίας δεδομένων. Κάποιες φορές είναι οι πάροχοι των υπηρεσιών και ε, αυτοί οι ίδιοι που επεξεργάζονται και τα στοιχεία ή αλλιώς ε, υπεργολαβικά κάνουν την επεξεργασία των στοιχείων. Θα πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν την διάκριση και τον καθορισμό του ρόλου του καθενός όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ε, γίνεται σεβαστό το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί το μήνυμα για όλους τους φορείς που θα πρέπει να υιοθετήσουν διάφορα κείμενα που ε, παραπέμπουν στις ίδιες έννοιες ενώ δεν αναφέρονται στις ίδιες πραγματικότητες και έχουμε και μια ολόκληρη κατηγορία δεδομένων και κριτηρίων για να έχουμε πρόσβαση στις διάφορες κατηγορίες δεδομένων και διατυπώνουμε αυτές τις ε, παρατηρήσεις για τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Νομολογίας για τα θέματα αυτά και για τους κινδύνους μιας αντίστροφης ερμηνείας των απαιτήσεων του δικαστηρίου για ορισμένες κατηγορίες δεδομένων που θα κατάλληλα για να, έχουμε λιγότερο προστατευμένα δεδομένα γιατί θα θεωρούνται λιγότερο ευαίσθητα μείνει έτσι ως έχει αυτή η πρόταση. Γιατί για τα στοιχεία των συνδρομητών ή τα στοιχεία της πρόσβαση οι εγγύσεις είναι λιγότερο σημαντικές από αυτές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή για τα, δικαιο... για τα στοιχεία δεδομένων ή συναλλαγών. Τα τελευταία μας σχόλια αφορούν την ίδια διαδικασία και τις διάφορες, τα διάφορα στάδια αυτής και σημεία για τα οποία θα επιθυμούσαμε επιπλέον εγγυήσεις. Καταρχάς για το αρκετά χαμηλό κατόφλι που επιτρέπει να εκδοθούν εντάλματα. Ήδη έγινε αναφορά στην έλλειψη εναρμόνισης του ποινικού δικαίου μέσα στην Ένωση και το γεγονός ότι ορισμένα εντάλματα, για ορισμένα εντάλματα μάλλον το γεγονός ότι είναι ποινικό αδίκημα αρκεί, ενώ αλλιώς ε, σε κάποια άλλα υπάρχουν ε, ανώτατες ποινές τριών ετών αρκετά χαμηλά κατόφλια δηλαδή που καλύπτουν σχεδόν όλα τα δικήματα. Έπειτα, πιο σύντομε προθεσμίε για την ε, υποβολή των δεδομένων. Μπορεί να υπάρχει ένα κριτήριο ανάγκη. Όντω, δηλαδή εκεί θα πρέπει να υποβληθούν ε, πιο σύντομα τα δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πλήρη έλλειψη των εγγύσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν posteriori να ελέγχονται τα στοιχεία και του κατά πόσο έγιναν σεβαστές οι διάφορες διαδικασίες. Τρίτη σειρά παρατηρήσεων αφορά το, που αφορούν το, θέμα των εγγυήσεων που θα μπορούσαν να προβλεφθούν ώστε να μην υπάρξουν καταχρήσεις, ας πούμε η συσχέτιση ανάμεσα στη διαδικασία διατήρησης και υποβολής των δεδομένων που αυτά τα δύο δεν συνδέονται απόλυτα πάντα. Τη στιγμή που έχουν παγώσει τα δεδομένα, ας πούμε, η εντολή παγώματος των δεδομένων και το ένταλμα δεν είναι το ίδιο ε, ενώ η εντολή διατήρησης των δεδομένων δεν θα πρέπει να παραβαίνει ε, τη διάρκεια διατήρησης αυτών. Υπάρχουν μια ολόκληρη σειρά παρατηρήσεις για την ενημέρωση των αρχών προστασίας ε, των ενδιαφερόμενων ανθρώπων, ε, μεταφορά και εξασφάλιση αυτής. Οι τελευταίες παρατηρήσεις είναι ίσως οι πιο σημαντικές γιατί αφορούν τις διαδικασίες που επιτρέπουν να αντιστοιχούν να, να, να αντισταθεί κανείς στην εκτέλεση του εντάλματος. Η διαδικασία του άρθρου 14, δηλαδή η δυνατότητα του φορέα να αντιτεθεί στην υποβολή των δεδομένων όταν διαπιστώνουν σύγκρουση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων χαιρετίζει το γεγονός ότι προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Όμως το κατόφλι είναι αρκετά χαμηλό. Ένα ευρύτερο κατόφλι θα επέτρεπε να έχουμε έλεγχο πιο αποδοτικό όταν υπάρχουν ε, αντιφάσεις στο δίκαιο ή συγκρούσεις ε, δικαίου και επί τα δυνατότητα διαλόγου ανάμεσα στις ε, ευρωπαϊκές αρχές και τις αρχές τρίτων χωρών. Πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό. Για την ώρα όμως είναι πολύ στενά τα πλαίσια. Θα έπρεπε ίσως αυτό να προβλεφθεί σε περισσότερες περιπτώσεις ώστε να έχουμε μια εκτίμηση του Ευρωπαίου δικαστή ή, μπας περιπτώσει, των ευρωπαϊκών αρχών που θα πρέπει να βασίζονται, να βασίζεται μάλλον σε στοιχεία που να μην είναι πολύ απομακρυσμένα από τα πραγματικά στοιχεία που θα επιτρέπουν ένα διάλογο πιο τακτικό και πιο ε, ουσιαστικό. Σε αυτά θα σταματήσω γιατί τελείωσε ο χρόνος μου και νομίζω πως κάλυψα τις παρατηρήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω συνάδελφοι και όλοι οι προσκεκλημένοι μας κατανοούμε ότι ε, είναι μακρό το απόγευμα αυτό. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2.30. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας και να τονίσω ότι Όταν μιλάμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το, θέμα δεν αφορά μόνο την ε, προστασία των δεδομένων αυτό καθ' αυτό, αλλά μιλάμε για την προστασία των ίδιων των πολιτών. Γι' αυτό και είναι πάντοτε πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο τι είναι πραγματικά αναγκαίο στις, για τις έρευνες, αλλά ταυτόχρονα θα, θα προστατεύει και τους πολίτες μας, ιδίως τους ευάλωτους. Γι' αυτό και νομίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα τροφοδοτήσει και τις περαιτέρω συζητήσεις που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Κορνέλια, πολύ σύντομα. Με βάση τα όσα μας είπε η κυρία Μπρουνέ, έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι αρκετά στρόγγυλα, αν θέλετε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο κανονισμός, με δεδομένα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, μπορεί να βοηθήσει, έχει κάποια προστιθέμενη αξία. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, Ποια θα ήταν ενδεχομένω η εναλλακτική που θα μπορούσατε να προτείνετε στην Κομισιόν για να επιταχυνθούν διαδικασίε, για να καταστούν πιο αποτελεσματικέ οι διαδικασίε ή ισχύουσε. Ευχαριστούμε πολύ, Κορνέλια. Πολύ σύντομο ήταν το ερώτημά σου. Δεν ξέρω αν η απάντηση μπορεί να είναι εξίσου σύντομη. Κυρία Μπρουνέ, θέλετε να προσπαθήσετε τουλάχιστον να απαντήσετε. Σα ευχαριστώ. Είναι δύσκολο για τι αρχέ προστασία των δεδομένων να παρέχουν την ίδια σφαιρική ανάλυση όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άποψη τη προστασία των δεδομένων πρέπει να εξετάσουμε αν το, οι εγγυήσει είναι συμβατέ. Αυτό είπε και ο εκπρόσωπο του ελεγκτή των ε, δεδομένων. Γι' αυτό και από την άποψη της προστασίας των δεμένων θέλουμε όλα αυτά να είναι συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και, τη, και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όσον αφορά τις συστάσεις για να βελτιωθούν τα πράγματα, μία από τις γενικές συστάσεις είναι καλύτερα να αξιολογηθεί και να δοθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα υφιστάμενα μέσα δεν αποδίδουν. Είναι δύσκολο να σας πω τι θα πρέπει να βελτιώσουμε μέσα στο πλαίσιο άλλων οργάνων. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να γίνει κατά πρώτο λόγο, αλλά αυτό που προτείνουμε για παράδειγμα είναι η διαδικασία παγώματος των δεδομένων που φαίνεται να είναι ένας από τους λόγους που αιτιολογεί την ύπαρξη νέου μέσου, γιατί η πτυτικότητα των στοιχείων σημαίνει πως κάποιες φορές μπορεί να εξαφανιστούν τα στοιχεία πριν να τα έχουμε καν ε, μπορέσει να τα βρούμε. Εγώ ως αρχή λοιπόν προστασίας των δεδομένων κάπως δυσκολεύομαι να σας κάνω πιο συνολικές συστάσεις όσον αφορά το ποινικό δίκαιο ε, ή να αποδείξω ότι υπάρχουν δυσκολίες στα υφιστάμενα και προβλήματα στα υφιστάμενα και ισχύοντα μέσα. Πάντως, όπως είπα, εξ αρχής θα πρέπει να αποδειχτεί πως τα υπάρχοντα μέσα δεν λειτουργούν. Μία φράση. Για το παράδειγμα, ε, σε σχέση με τα όσα λείπουν ενδεχομένω. Λείπει, για παράδειγμα, η δυνατότητα να αξιολογήσει κανείς και να κατανοήσει την γνησιότητα μιας εντολής και των πιστοποιήσεων που συνοδεύουν τις εντελές από την χώρα έκδοσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ελέγχων που είναι ταυτόχρονα η εταιρεία που λαμβάνει και ε, αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά να διαπιστώνει ε, τον, το, τη γνησιότητα ε, της εντολής που έχει παραλάβει. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Αυτό που κρατάμε από το πάνελ αυτό είναι όχι μόνο η σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωτών δικαιωμάτων, αλλά ε, κυρίως από τις απαντήσεις που λάβαμε στο τελευταίο ερώτημα. Στο παρελθόν είχαμε αποφασίσει ότι όλα τα μέτρα για τις αστυνομικές και διοκτικές αρχές θα πρέπει να είναι περιορισμένα και στοχοθετημένα. Δεν υπάρχει ένας ε, τρόπο για να χειριστεί κανείς τις διαφορετικές υποθέσεις. Αυτό είναι μια κοινοτομία της νέας πρότασης όπου προτείνεται να θεσπιστεί μία νομική πράξη η οποία θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Ίσως λοιπόν θα ήταν ε, εύλογο να γίνει μια συζήτηση για την εξειδίκευση, την στοχοθέτηση των μέσων που θα θεσπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται στην πλειάδα των ε, ειδικών υποπεριπτώσεων που υπάρχουν ε, ε, στον, στις ένομες τάξεις της χώρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπόσνιακ, τον δικαστή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παρακολούθησε τη συζήτησή μας από το Στρασβούργο. Νομίζω ότι η όλη συζήτηση τροφοδότησε και την περαιτέρω συζήτηση που θα γίνει. Περνάμε απευθείας στο επόμενο πάνελ και καλώ τους ε, ομιλητές που έχουμε προσκαλέσει για αυτόν τον τελευταίο γύρο συζητήσεων, το τελευταίο τμήμα αυτής της σημερινής μας ακρόασης. Οι επόμενοι τρεις ομιλητές θα μας μιλήσουν για τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών, των ε, παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και καλούμε την κυρία Ελένη Κυριακίδου από την EPIC, την Λόρα Βάγνερ από τη Vodafone και τον δόκτορα Μαξιμίλιαν Σούμπερ που είναι αντιπρόεδρος της EuroISPA. Σας καλωσορίζω και όπως ε, και όλοι οι άλλοι ομιλητές έχετε περίπου 8 με 10 λεπτά για να μας κάνετε τις παρουσιάσεις σας και ξεκινάμε απευθείας με την Ελένη Κυριακίδου από την EPIC στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που με απίφθινε. Είμαι η Ελένη Κυριακίδες, είμαι ε, ε εργαζόμενοι στην EPIC που είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό την παρακολούθηση ζητημάτων που σχετίζονται με θεμελιώδη δικαιώματα ατομικές ελευθερίες. Θα σας παρουσιάσω τις δικές μας συστάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις διασυνοριακές περιπτώσεις. Υπάρχουν ένομα συμφέροντα των διεκτικών αρχών να λαμβάνουν δεδομένα σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον. Ωστόσο, αυτή η ανάγκη ε, δημιουργεί την ανάγκη να υπάρχουν εχέγγυα για τις ατομικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε συλλέξει ως εμπειρία στις ΕΠΑ. Η είπα, ε, θέσπισαν το δικό τους ε, ρυθμιστικό πλαίσιο έπειτα από αποφάσεις ε, των δικαστηρίων μας. Στην περίπτωση Ηνωμένες στην υπόθεση υπόθεση ε, Ηνωμένες Πολιτείες έναντι, κατά της Microsoft ε, απαχωρε, επετράπει αρχές να, υποχρεώσουν τη Microsoft να, παραδώσουν, να παραδώσει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα χρηστών. Ε, ταυτόχρονα θεσπίστηκαν διάφορες ε, προδιαγραφές για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, δύο στοιχεία ήταν τα βασικά της, ε, της απόφασης του δικαστηρίου. Αφενός, τροποποιήθηκε η, η οδηγία ε, υποχρεώνοντας τους παρόχους να διατηρούν τα δεδομένα είτε τα αποθηκεύουν εντός είτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα να, ε, οι, πάροχοι να προσφεύγουν κατά της απόφασης και αυτή, δίνεται, ε, αυτή δίνεται, δίνεται μόνο όταν υπάρχει αντίθεση, ή σύγκρουση νομοθεσίας και όταν υπάρχει εκτελεστική απόφαση, εκτελεστική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και ε, νομοθεσία που προβλέπει παρόμοιες δυνατότητες για, ε, όπως αυτές που προβλέπονται στις ΗΠΑ. Επίσης, ε, δίνεται δυνατότητα σε εξωματούχους των ΗΠΑ να ε, ε, ζητούν την παρακολούθηση και την αποθήκευση δεδομένων. Έπειτα από από μια, τη λήψη μια τέτοιας απόφασης πρέπει γραπτός το Κογκρέσο να εγκρίνει ε, μια τέτοια διαδικασία και να τηρούνται τέσσερα κριτήρια. Τα κριτήρια ε, αυτά τα τέσσερα είναι τα εξής. Πρώτον, η ένομη τάξη της ε, αλλοδαπής της ξένης χώρας θα πρέπει να, ε, έχουν, να, έχει να έχει επαρκή στοιχεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ξένη κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να ε, έχει λάβει μέτρα σχετικά με τη διάδοση πληροφοριών που αφορούν Αμερικανούς πολίτες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να, να αποκρυπτογραφούν ε, προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να πληρούνται κάποιε συγκεκριμένε προποθέσει όσον αφορά την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων των Αμερικανών πολιτών. Ε, μια σειρά από εχέγγυα για εντολέ και συμμόρφωση. Αν το Κογκρέσο δεν εκφράσει εντός 180 ημερών την αντίρρησή του, τότε ε, αναλαμβάνεται δράση αυτεπάγγελτα. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού Οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης ΕΠΙΚ έχουν ασκήσει δρυμία κριτική κατά αυτού του συστήματος. Σε ένα σύστημα μονο, μονόπλευρης ε, πρόσβασης, όταν μια χώρα μπορεί να μην γνωρίζει καν ότι έχει υπάρξει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα, πόσο μάλλον να μπορεί και να ε, μπλοκάρει τέτοιες, ε, τέτοια πρόσβαση, χρειάζεται να διαπιστώσει κανείς ότι παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα. Ακόμη και σε χώρες όπου υπάρχουν ε, εύρωστοι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορούν να παραβιαστούν αυτά ε, μέσα αυτών των διαδικασιών. Σε χώρες όπου δεν υπάρχουν ε, νομικά εχέγγυα και ε, ισχυρή ε, νομοθεσία, τα, προ... τα προβλήματα αυτά θα είναι ακόμα ισχυρότερα. Ως αποτέλεσμα, αν θεσπιστούν μέτρα άμεσης πρόσβασης θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ύψιστα δυνατά εχέγγυα. Και εδώ θέλω να έρθω στις συστάσεις μας για τις προτάσεις για τη δυσενορική πρόσβαση. Πρώτον, πρέπει να απαιτούνται ε, νομικά προστατευτικά εχέγγυα για, την προσωπικά, τα προσωπικά δεδομένα ε, στις διασυνορικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένε απαιτήσει για την κοινοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων και ανομοποίηση όλων των άλλων στοιχείων που δεν σχετίζονται με την έρευνα. Δικαστική αναθεώρηση που είναι το καλύτερο ένδικο μέσο θα πρέπει να προβλέπετε επίσης η και επίσης συστήνει την ε, έγκριση ε, πρόσθετων εγγυήσεων που θα αντισταθμίζουν τη μονομερή διάσταση ε, αυτών των εντολών. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα κόστος το οποίο επομίζεται τρίτη χώρα, τότε μπορεί να χρησιμοποιείται έμλατ Επίση, θα πρέπει αυτέ οι υποθέσει να αφορούν μόνο περιπτώσει όπου έχουν διαπραγματευτεί πράξει που είναι αξιόπινε και υπό τι δύο εθνικέ ε, ένομε τάξει. Για να εξασφαλιστεί ότι ε, η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται μόνο όπου είναι απολύτω απαραίτητο. Θα πρέπει να υπάρχουν επίση μέσα προσφυγή. Για παράδειγμα, Πιστεύουμε ότι οι ΙΠΑ μπορούν να ξεκαθαρίσουν ποια είναι τα ένδικα μέσα για μη Αμερικανούς πολίτες, των οποίων τα δεδομένων έχουν τύχη πρόσβασης από ε, τρίτες χώρες, τρίτους φορείς. Για παράδειγμα, όπως η πρόταση e-evidence, η EPIC ε, συστήνει να προκρίνεται η εντολή διατήρησης στοιχείων όταν, δεν μπορεί, όταν η, η εντολή υποβολής στοιχείων δεν πληρεί όλα τα κριτήρια. Αυτό μπορεί να εμποδίσει συγκεκριμένες μη νόμιμες, αν θέλετε, εντολές έως ότου ξεκαθαριστεί η πορεία των ερευνών. Επίσης, απαραίτητη είναι η καταγραφή ε, λεπτομερών στοιχείων για τον αριθμό και το είδος των εντολών που εκδίδονται. Οι εκθέσεις Wired από τον ΙΠΑ, ε, για παράδειγμα, ε, οδήγησαν στην εξειδίκευση και την τροποποίηση της Αμερικανικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Θέση μας είναι ότι ανεξάρτητα από τον ε, μηχανισμό επιβολής του νόμου θα πρέπει ε, αυτό να εξασφαλίζεται στο ύψιστο δυνατό επίπεδο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας σήμερα και είμαι στη διάθεση για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα άκουσα με προσοχή και άκουσα σε πολλέ περιπτώσει τη λέξη δικλίδα ασφαλεία, ε, τη λέξη ένδικα μέσα. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο νομικό εργαλείο, τέτοιες δικλείδε ασφαλεία και ένδικα μέσα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζουν οι αρχές, ε, όχι οι ιδιωτικοί φορείς. Να περάσουμε στον επόμενο μιλητή μας, την επόμενη ομιλητρία μας, ε, η κυρία της Λαουρά Βάγκανερ από τη Vodafone. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ανέβει η παρουσίασή μου στην οθόνη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ε, προσκαλέσατε, που προσκαλέσατε την Vodafone. Χαιρόμαστε που μπορούμε να δώσουμε και την προοπτική ενός παρόχου, γιατί αναφέρθηκαν προφανώς πολλοί παρόχοι σήμερα το απόγευμα. Είναι πολύ ευρία πολύ ευρύς ορισμός τους ε, στην πρόταση. Ποιοι είμαστε λοιπόν και περιμένω να δω και τις διαφάνειές μου. I know. you don't think you might start without? Uh, yes, I can. I can. If you bring up the second slide as I go through, I also have a USB stick. If uh, we go to. Αν θέλετε να περάσω κατευθείαν στη δεύτερη διαφάνεια, το έχω και σε USB stick την παρουσίαση. Λέει η κυρία Βάγκνερ, είμαστε μια παγκόσμια λοιπόν εταιρεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως ε, εθνικές ε, άδειε και ρυθμιζόμαστε από τις εθνικές ε, νομικές πραγματικότητες. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη μας αγορά, η Μάλτα η πιο μικρή μας αγορά. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα σύγκριση των νομοθεσιών σε ό,τι αφορά το έγκλημα και την έρευνα για τα εγκλήματα, τις ποινικές ερευνές. Πάντα λοιπόν δρούμε με άδειε σύμφωνα με του σχετικού κανόνε για τι τηλεπικοινωνίε. Αυτό σε ό,τι αφορά του παρόχου και η άδειά μα περιλαμβάνει υποχρέωση συνεργασία με τι εθνικέ αρχέ επιβολή του νόμου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν δεν συνεργαζόμαστε, δεν συμμορφούμαστε με τον νόμο και μα αφαιρείται η άδεια. Είναι σημαντικό αυτό γιατί αυτό δεν ισχύει για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που καλύπτονται από την πρόταση αυτή. Δεύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη δέσμευση για την ε, προστασία των καταναλωτών μας και των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό είναι τμήμα της άδειά μας. Αν δεν μας ε, εμπιστεύεται οι καταναλωτές, αυτό υπονομεύει τον όγκο της ε, εργασίας μας. Also mentions that we have... Η διαφάνεια αναφέρει ότι Okay. Um, so we have um, a long-standing experience. Έχουμε μακρά λοιπόν εμπειρία σε ό,τι αφορά τέτοιες υποχρεωτικές διατάξεις, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα από τις αρχές υποβολής του νόμου και αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προστατεύσουμε το κοινό και να ε, βοηθήσουμε τις αρχές ε, προστασίας ε, του νόμου. Να σας πω που είναι η διαφάνεια, η παρουσίασή μου. There. There. Thank you. Sorry, everyone. Um, It's just going to be easier for all of us if we also have some. Θα είναι λίγο πιο απλό αν έχουμε και την παρουσίαση στη διαφάνεια να την παρακολουθήσουμε. So voilà, just to make the, the point again, refusal to comply in our national context where we do cooperate with law. Η άρνηση συμμόρφωσης δεν σημαίνει um, έγκριση Όλα αυτά λοιπόν που θα σας πούμε δεν βασίζονται, δεν τα βγάζουμε από τον αέρα. Προσπαθήσαμε να είμαστε πάντα διαφανείς σε ό,τι αφορά τις εντολές που λαμβάνουμε. Δεν είναι πάντα υποχρεωτική το αίτημα αυτό. Θεωρούμε ότι αυτό αποκαλύπτουμε τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις χώρε τι οποίε δραστηριοποιούμαστε. Αυτό προφανώς είναι πολύ διαφορετικό. Και είναι συνεκτικό, καλύπτει πολλά πράγματα και αν θέλετε να το διαβάσουμε. Τρίτη διαφάνεια. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να κρατάμε τέτοια δεδομένα, κάνουμε επεξεργασία τέτοιων μετατέτα, οποιαδήποτε τέτοια βελτίωση και γίνεται διάφορε συζητήσει στο Συμβούλιο, δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο για τα δεδομένα περιεχομένου. Δεν επιτρέπουμε λοιπόν τέτοια πρόσβαση εκτός και αν υπάρχει τέτοια νομική προδιαγραφή, δεν δίνουμε τελούσια τέτοια στοιχεία για τους πελάτες μας. Αυτό συνάδει και με αυτά που ανέφερα προηγουμένω σε ό,τι αφορά την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε εντολή ε, από αρχή εκτός δικαιοδοσίας της, δηλαδή αποδεχόμαστε τις εντολές μόνο από τις αρμόδιες αρχές και οι, τα αιτήματα από αλλαδαπές αρχές δεν είναι κάτι στο οποίο ανταποκρινόμαστε τώρα. Επίσης δεν αξιολογούμε τον σκοπό, την πρόθεση οποιασδήποτε τέτοια εντολής. Όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο τα επεξεργαζόμαστε με λίγες ή μηδαμινές πληροφορίες σε ό,τι αφορά το υπόβαθρο του αιτήματο. Αυτό για μας ως πάροχος, ως εταιρεία τηλεπικοινωνιών δεν μας αφορά όπου τίθεται θέμα μη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία και με τις τυπικές διαδικασίες δεν είναι ε, δυνατόν και ούτε καν ευκταίο να αξιολογήσουμε το υπόβαθρο της ε, εντολής που μας υποβάλλεται. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι δεν είμαστε αντίθετοι επί της αρχής σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή. Αυτό που βλέπετε στην παρουσίασή μου είναι ότι θα λειτουργήσει το σύστημα μόνο αν είναι ξεκάθαρα ποιο κάνει τι και θα αντιευκρινιστεί αυτό το κομμάτι. Επόμενη διαφάνεια. Τι συζητάμε λοιπόν σήμερα, ποιο είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση κατέδειξε που βρίσκεται το επίκεντρο των ζητημάτων και ο κύριος Κέρκοφ και οι υπόλοιποι πριν από μένα αναφέρθηκαν επανελειμμένα σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία τα οποία τους δυσαρεστούν ε, σε ό,τι αφορά τις εταιρείε που δεν είναι στην παρούσα φάση υπό ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Και εδώ βλέπετε ένα απόσπασμα από τις ε, συχνές ερωτοπαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βελτιωθεί η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά τεκμήρια. Κάποιες από αυτές τις εταιρείε λοιπόν δεν υπάγονται σε αντίθεση με εμάς σε εθνικές δικαιοδοσίες και θα ήθελα να το σκεφτείτε παρακαλώ αυτό Θέλουμε εδώ να υπάρξει αναλογικότητα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό για τους παροχούς. Μέσα σε έξι ώρες ε, το χρονικό διάστημα εκτέλεση ανάγκη. Αυτό θα πρέπει να μας, είμαστε έτοιμοι. Για αυτό το διάστημα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ε, εντολή αυτή εδώ, στον κανονισμό, στην πρόταση μάλλον. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δεκλήτα ασφαλεία που μας επιτρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Το ποιο ζητάει τι. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας ε, αναφέρει το πώς θα πρέπει να αποκαλύπτονται τα στοιχεία μέσω ασφαλών πλατφόρμων, θα προτιμούσαμε ιδανικά να υπάρξει μια κεντρική πλατφόρμα με σαφείς ελέγχου πρόσβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν διευκρινίσουμε το πώ πρέπει να χορηγούνται τα στοιχεία αυτά, κατά πάσα πιθανότητα θα λάβουμε τέτοιε εντολέ χαμηλής ποιότητα και αυτό θα υπονομεύσει όλη τη διαδικασία και του σκοπού τη πρόταση. Μας ε, ζητείτε να κάνουμε έναν έλεγχο νομιμότητας ε, και αναλογικότητα. Αυτό που κάνουμε είναι ελέγχου σε ό,τι αφορά την τήρηση των τυπικών διαδικασιών. Αυτό δεν είναι... έχει να κάνει με τις επίσημες ε, εγκεκριμένε αρχές που... Αλλά δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ελέγχουμε το υπόβαθρο μια εντολή την οποία λαμβάνουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε κατά πόσον βάση των στοιχείων αυτών θα αποκαλύπτουμε ή όχι τα στοιχεία δεν αισθανόμαστε ότι είναι δικό μας ο ρόλος αυτός. Για θέματα ευθύνη. Αυτό αναφέρθηκε εν συντομία και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αν είμαστε, αν συμμορφούμαστε, φύγετε με τις υποχρεώσεις για τα ηλεκτρονικά τεκμηρία, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι σε ό,τι αφορά τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Εδώ τίθεται ένα θέμα για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια και το GPDR. Αν ένας πάροχος υπηρεσιών συμμορφούται με τα τεκμήρια και υποχρεούμαστε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία ενός καταναλωτή, θα πρέπει να υπάρχει διευκρίνηση ότι αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 23 του GDPR. Αυτό λοιπόν είναι ύψιστη σημασία για μας. Γιατί αυτό θα καθόριζε την αποτελεσματικότητα της πρότασης. Ένα σημαντικό σημείο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε. Το θέμα του αντικτύπου κόστους. Η αρχική πρότασή μας δεν συγκεκριμένο ρόλο σε ό,τι αφορά το φόρτο εργασία. Βλέπετε στην διαφάνεια ότι είμαστε μεγάλο πάροχο. Χρειάζεται να έχουμε διαρκώ ε, έτοιμε ομάδες για όλα τα βήματα τα οποία σα ήδη περιέγραψα. Σας ήδη. Αν προβλέπετε ένα ευρωπαϊκό διαστοριακό σύστημα για τη βελτίωση της πρόσβασης ε, των δεδομένων στα δεδομένα, θα πρέπει κατελάχιστον να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής. Άρα αυτοί οι κανόνες είναι από λειτουργικής άποψης. Όσο πιο πολύ ε, είναι σε λειτουργικό επίπεδο οι κανόνες, όσο πιο ξεκάθαρα θα δίνεται πράγματα για τους παρόχους. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε ότι η αποκάλυψη δεδομένων δεν γίνεται σε ένα κλικ. Υπάρχει και το στοιχείο του κόστους. Χρειαζόμαστε τέσσερις ομάδες. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την εντολή, να κοιτάξουμε και τα δεδομένα. Όχι μόνο την εντολή, αλλά και τα δεδομένα. Να τεκμηριώσουμε κάθε βήμα της διαδικασίας την εντολή, την εξαγωγή των δεδομένων, την αποκάλυψη. Αυτό καθορίζει τι μετα χρειαζόμαστε. Να τα εξετάζουμε αν στέκουν. Ενδεχομένω να χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή με τι ε, αρμοδίε αρχέ σε περίπτωση που κάτι είναι ασαφέ. Επικοινωνία, μετάφραση τη επικοινωνία. Αυτό δεν προβλέπεται. Το κόστο από την ε, πρόταση. Μετά κάνουμε την εξαγωγή βάσει των metadata Κάνουμε παλήθευση, εξασφαλίζουμε ότι είναι ασφαλή και μόνο τότε αποκαλύπτουμε και ελέγχουμε αν πληρούνται όλα τα πρότυπα σε διαφορετικά αφορά τα τεκμήρια, όπω προβλέπονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα όλα αυτά θα γίνουν ε, γρήγορα. Αλλά τίποτα στην πρόταση δεν εξασφαλίζει ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Μιλάμε για 27 αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που αναμένουμε εμείς είναι αύξηση των εντολών και των ετοιμάτων. Στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή είναι η μοναδική ωραία εικόνα που έχω στην ε, διαφάνειά μου σε σύγκριση και με τους προηγούμενους ε, ομιλητές. Να σας παρουσιάσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για να σας δείξω πόσο περίπλοκη και επισφαλής είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς ως παροχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές. Ε, οι πιο πολλές υποθέσεις είναι ασφαλείς, οριακές. παραδείγματα ενδεχομένων εγκλημάτων. Υπάρχει η προστασία των πηγών για του δημοσιογράφου. Τι γίνεται αν ένα δημοσιογράφο είναι σε μια ξένη πρωτεύουσα και είναι αντικείμενο έρευνας από κάποιες αρχές. Οι αρχέ, η νομοθεσία για την προστασία των πηγών είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα. Ποιος αποφασίζει τι. Η άμβλωση είναι έγκλημα σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες όχι. Εμείς ως πάροχος θα εξεθούμε, θα αναλάβουμε την ευθύνη. Αν παρέχουμε δεδομένα, γιατί πολύ απλά πρέπει να τηρήσουμε τις νομικές προδιαγραφές και το θέμα της προστασίας των παιδιών. Τι είναι η ηλικία συνένεση, ποιο είναι ενήλικο ή για παράδειγμα οι ομιλίε μίσου Για να σας δώσω κάποια πράγματα να σκεφτείτε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε ούτε θέλουμε να είμαστε νομικοί οι δήμονες σε τέτοια θέματα. Πόσο μάλλον που αυτό αφορά και 27 διαφορετικές χώρες μέλη με διαφορετικά συστήματα. Εμείς είμαστε ειδικοί σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, σε ηλεκτρονικά συστήματα. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Και εδώ πάμε στη τελευταία μου διαφάνεια. Θα περιοριστώ πλέον σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα θα επιληθούν αν ε, εγγυηθούμε την ε, αυθεντικότητα του αρχών, έλεγχος νομιμότητας, οι αρχές γνωρίζουν καλύτερα από όλους ε, το νομικό του σύστημα. Αυτή είναι η δουλειά τους και επιστροφή κόστος σε ό,τι αφορά το εθνικό πλαίσιο. Οι εθνικές αρχές επίσης θα πρέπει να ασκήσουν τις αρμοδιότητες επικυριαρχίας τους, όχι οι υπάροχοι στη λειτουργική διάσταση έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε να επανεφεύρουμε από τεχνική άποψη τον τροχό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη εντολή αυτή. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίηση έχει ω καθήκον να επιλύσει τέτοια συστήματα ισοτιμία μεταξύ των εθνικών συστημάτων και εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί για όλου. Πολλή δουλειά λοιπόν ήδη γίνεται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του EIO και αυτό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε ό,τι αφορά και τα τεκμηρία αυτά. Θα σας ευχαριστήσω λοιπόν που με ακούσατε και την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κατά κάποιο τρόπο κάπως ε, ιδιωτικοποιείται το ποινικό δίκαιο από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον στι επιπλέον ε, συνεδριάσει με τον εισηγητή και τους Κιώδης. Έχουμε το τελευταίο μιλητό, το Μαξιμίλη Σούπερ, που είναι αντιπρόεδρος του κ. ΕΣΠ. Δεν ακούγεται ο μιλητή. Ναι, καλύτερα είναι να ανάψω και το μικρόφωνο μου, λέει ο μιλητή. Καταρχά σα ευχαριστώ που με καλέσατε για να εξηγήσω ε, τι απόψει τη Ευρωπαϊκή. Ε, Βιομηχανία του ίντερνετ για αυτό το σημαντικό θέμα και εγώ περιμένω Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και προσπάθησα να τις δείξω με βάση την άποψη της βιομηχανίας. Μιλάμε για ένα σύστημα ανταλλαγή δεδομένων που όχι μόνο θα περιορίζεται στις κατηγορίες ε, δεδομένων για τις οποίες μιλάμε σήμερα ε, είναι προφανές για τους περισσότερους ότι αργά ή γρήγορα αυτό το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους, ας πούμε για την ε, ε, σύλληψη σε πραγματικό χρόνο, για τις τράπεζες κτλ. κτλ. Άρα θα πρέπει να αναπτύξουμε κάτι που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι όμως όταν το κάνουμε αυτό και να λάβουμε υπόψη ενδεχόμενα που μπορεί να αποδεχτούν προβληματικά για να προσπαθήσουμε εκ των προτέρων να τα αποφύγουμε. Επόμενη διαφάνεια. Όταν μιλάμε για το Euro ΕΣΠΑ, ε, ε, το αρχίσαμε πριν από 20 χρόνια. Ε, όμως ε, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε πολύ μεγάλο εύρος μελών και άρα μελετούμε διάφορα νομικά συστήματα. Έχουμε 2.500 περίπου εταιρείε, οι οποίε είναι οι περισσότερε μικρομεσαίε και θα επανέλθω σε αυτέ ε, στην παρουσίασή μου. Είναι οι χαρακτηριστικές εταιρείε ISP που ε, απασχολούν 3 με 10 υπαλλήλου. Το να μιλάμε για προθεσμίες, υποχρεώσεις για όλους αυτούς είναι κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Η εισήγησή μου ίσως είναι καλή για να κλείσουμε αυτήν την ημέρα, γιατί θα συνοψίσω κάπως τα όσα υπόθηκαν σήμερα. Ε, επιβολή ε, ε υποβολή στοιχείων από μια εταιρεία. Τα στοιχεία πάνε και έρχονται. Οπότε αν το δούμε από την άποψη μιας τρίτη χώρας βλέπουμε ότι αυτή η σημερινή διαδικασία ΕΜΛΑΤ είναι πολύ περίπλοκη γιατί ε, συμμετέχουν ένα σωρό αρχές και συμφωνώ και με του ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε την ενδεχόμενη δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος ΕΜΛΑΤ. Ε, συμφωνούμε πως ε, είναι κάπως περίπλοκο. Ακόμα και αν ε, εξετάσουμε την Ευρώπη, για παράδειγμα, εξακολουθούν να, αναμεχνύονται πολλές ε, αρχές ε, και αν δούμε αυτή την πρόταση για ηλεκτρονικές αποδείξεις. Βλέπουμε την παραδοσιακή αρχή στο κράτος Β, που είναι το κράτος που λαμβάνει τα δεδομένα και τότε έχουμε το ερώτημα ποιος θα πρέπει να αντισταθμίσει τη δεύτερη αρχή που ε, θα εγγυηθεί την μεταφορά ή την επιστροφή που θα γίνει στο μέλλον. Uh, respect. Το γύρο ΙΣΠΑ έχει κάποιες απόψεις εδώ. Την πρώτη αφορά την έλλειψη ενσωματωμένων διαδικαστικών ε, εχεγγύων. Ένα κράτος εκδίδει την εντολή το δικαστήριο μάλλον εκδίδει την εντολή και αυτό το κάνει μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Θα πρέπει να εξασφαλίσει πως το ένταλμα το οποίο εκδίδει είναι αναλογικό και ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη ανεξάρτητη αρχή που θα κάνει τον έλεγχο αυτό και δεν θα εξαρτώμεθα μόνο από την πρώτη αρχή. Δεν θέλω να αφήσω καμία αφιβολία ότι ως μηχανία του ίντερνετ στηρίζουμε τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ωστόσο όπως εξηγήθηκε και με λεπτομέρειες προηγουμένως θα υπάρχει, θα είναι θετικό το να υπάρχει και ένας δεύτερος ανεξάρτητος έλεγχος για τα εντάλματα που εκδίδουν τα κράτη και γι' αυτό και ζητούμε την ύπαρξη μιας αρχής. Κάποια από τα μέλη μας θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν έναν επιπλέον έλεγχο για να ελέγξουν την ανάγκη και την αναλογικότητα, αλλά μην θεωρήσετε ότι θα είναι κάποιο, κάποια αποζημίωση θα είναι μια επιπλέον ε, ε, εγγύηση για τους προμηθευτές, ε, τους παρόχους ίντερνετ. Τώρα, όταν μιλάμε για το εγκληματικό κατόφλι, υπόθηκε προηγουμένως ότι αυτό κυμαίνεται ανάμεσα στα κρατημέλη, αλλά και ότι μπορεί να είναι εύκολο για τον νομοθέτη του κράτους μέλου να αυξήσει τα όρια. Όταν μιλάμε για κατόφλι, Μιλάμε για τα, τα, τα, τα δεδομένα περι, περιεχομένου, ενώ τα δεδομένα για τους συνδρομητές μπορεί να μην φτάνουν για να φτάσουν σε αυτό το κατόφλι. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει καμία εξαιρετικά ευρεία λίστα ή κατάλογος για το ποια αδικήματα θα διώκονται ή όχι και πώς. Πάλι δηλαδή εδώ έρχεται το, η δοκιμή αναγκαιότητας και αναλογικότητας που θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Ένα από τα θέματα που είναι βασικό είναι για τους ε, παρόχους υπηρεσιών Ιντερνετ είναι η αρχή της διπλής ε, κλιματικότητας. Αυτός είναι ένας ακρογωνιαίος λήθος ε, όταν διώκει κανείς σε κλίματα στο ίντερνετ. Θα πρέπει να προσέχουμε να μην το ξεχάσουμε γιατί παραμένει στον πυρήνα του ενδιαφέροντος ε, των παρόχων. Όταν μιλάμε για πρακτικούς στο δικό μας τομέα, αυτό είναι καθημερινή δουλειά. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, προβλέψεις ε, για σύγκρουση κανόνων ή νόμων. Το θέμα της ε, του ελέγχου της αυθεντικότητας του αιτήματο επίσης είναι σημαντικό και το ανέφεραν ε, πολλοί συνάδελφοι. Μπορεί ας πούμε να είναι ε, τρεις άνθρωποι στη μέση της Αυστρίας και να λαμβάνουν ένα ένταλμα από μια ξένη αρχή και θα είναι πολύ δύσκολο να να καλύψουν αν η εντολή στάλθηκε πραγματικά από κάποια πορτογαλική δικαστική αρχή ή από κάποιο γερμανικό αστυνομικό τμήμα στο μέλλον αδρυμό. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους ελέγχου της αυθεντικότητας της εντολής που μας φτάνει. Επίσης και λόγω του GDPR εμείς ως βιομηχανία έχουμε επενδύσει πόρους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οποτεδήποτε γίνεται μεταφορά δεδομένων μέσα στις εταιρείε μας και ανάμεσα στις εταιρείε μας να ε, ισχύουν συγκεκριμένα στάνταρ ασφάλειας και ακαιρεότητας. Και αυτό μας ε, οδηγεί στο να, στο να σκεφτούμε και τον ενδεχόμενο κίνδυνο όλα τα οι Internet Providers στην Ευρώπη, να χρειαστεί να μειώσουν τις προδιαγραφές ασφαλείας τους. Ας πούμε, αν αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε μηχανήματα fax στο μέλλον, ε, το οποίο σας διαβεβαιώ είναι εξαιρετικά προβληματικό, γιατί οι περισσότερες από τις εταιρείες μας δεν έχουν πια φάξ, ενώ στο δημόσιο τομέα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα φάξ. Ενιαία σημεία επαφής. Και αυτό θεωρήθηκε πολύ σημαντικό. Γιατί, γιατί όταν έχουμε ένα μόνο σημείο επαφής, από τεχνικής άποψη είναι πολύ πιο εύκολο να ανταλλαγούν ε, στοιχεία κρυπτογραφημένα γιατί έτσι θα, ανταλλαγούν πιο εύκολα και τα κλειδιά. Αλλά επίσης μπορεί να γίνει και ένας ποιοτικό έλεγχος πριν να σταλούν ε, όλα αυτά στον ε, πάροχο. Στην Αυστρία, ας πούμε, λάβαμε εντάλματα που λείπαν υπογραφές ή ε, απαραίτητες πληροφορίες. Ενώ όταν υπάρχει ένα μόνο σημείο επαφής, όπως έχει φτιαχτεί τώρα, αυτό σημαίνει ότι από την πλευρά του δημόσιου τομέα, το αίτημα που φτάνει στον ε, πάροχο είναι ομοιόμορφο. Και άρα ο χρόνος που θα χρειαστεί για την επεξεργασία του και για την παράδοσή του θα μειωθεί. Επόμενη διαφάνεια. You see uh, the potential downsides of a fax message and now just imagine you're receiving this from an uh, from a public authority who is missing uh, who is looking εδώ βλέπετε ένα ένταλμα για, από κάποια αρχή που ε, αναζητεί κάποιον άνθρωπο, κάποιον αγνοούμενο. Τι Εδώ, αυτή είναι η διαφάνεια που σας έλεγα. Αυτό φαίνεται. Τα φαξ είναι τεχνολογία του περασμένου αιώνα, της περασμένης χιλιετίας και δεν θα θέλαμε να την αναγκαστούμε να την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ε, δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε πια τα ίδια συστήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα στοιχεία εδώ περνάνε ανάμεσα στους παρόχους και στις αρχές επιβολής του νόμου. Εδώ η διερμηνία σταματά. Καλό σας βράδυ. Yes, when it uh, comes to notification, there are two scenarios. One of them is uh, notification to users. Here, as we, we are convinced that transparency should be the rule, uh, not confidentiality. When it comes to notification of judicial authorities, I think this is going into the right direction